Colleagues, can I call the meeting to order? You have before you the... Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνεδρία. Έχετε ενώπιόν σας την ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε με αυτήν? Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο είναι οι κατευθυντήρες γραμμές TNT, εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών. Δύο συγγητές είναι εδώ, ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος Έρτουγ. Οπότε, ποιος θα πάρει πρώτος το λόγο, Γιώργο, ο κύριος Κουμουτσάκος. Έχετε το λόγο κύριε Κουμουτσάκο. Ευχαριστώ, Μπράιν. Έως τώρα έχουμε κάνει τέσσερις συναντήσεις με τους σκιώδεις συζητητές. Θα σας δώσω μια γενική εικόνα του πού βρισκόμαστε. Ε, έχουμε κανονίσει ακόμα μία συνάντηση για αύριο με τους σκιώδης και προβλέπουμε να γίνει άλλη μία συνάντηση στο Στρασβούργο. Θέλω να πω σε όλους τους συναδέλφους ότι αν χρειαστεί και τρίτη μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπάρχει το οποίο θέλω να σεβαστούμε απολύτως, δηλαδή τη 18η Δεκεμβρίου ημέρα ψηφοφορίας. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρξει ανάγκη, θα κανονίσουμε και άλλη συνάντηση, τρίτη πέραν των δύο που ήδη προβλέπονται. Τώρα, όσον αφορά τις ε, συμβιβαστικέ προτάσεις. Έχουν κατατεθεί 22 συμβιβαστικές τροπολογίες που αφορούν σε 11 άρθρα ε, του σχεδίου κανονισμού. Έχουν κατατεθεί 11 συμβιβαστικές ε, προτάσεις που αφορούν recitals και 19 συμβιβαστικές προτάσεις που αφορούν στα παραρτήματα και τους χάρτες. Ε, σύνολο περίπου 50-52. Μένουν ακόμα εκκρεμή ορισμένα θέματα και τις αμέσως επόμενες μέρες θα προσθεθούν ακόμα μερικές συμβιβαστικές προτάσεις, αλλά λίγες. Μέχρι στιγμής έχουμε συζητήσει, πιστεύω, εξαντλητικά και με καλή διάθεση και επικοδομητικό πνεύμα συμβιβαστικές προτάσεις που αφορούν τα ακόλουθα άρθρα. Το άρθρο 3 που αφορά θα τα πω στα αγγλικά, Definition on European Added Value. Article 3, Definition on Cross-Border Section. Άρθρο 3, καθορισμός για τις ε, διασυνοριακές τομές. Άρθρο 3, ορισμός για τις αστικές ε, καταστάσεις. Άρθρο 4, ε, στη, στόχοι. Άρθρο 5, επίσημο δίκτυο. Άρθρο 10, προτεραιότητες. Άρθρο 12, στοιχεία υποδομών. Άρθρο 16, παράγραφος τρία Συνδεδεμένοι εξοπλισμοί για πλωτούς, πλωτές οδούς <clears throat> εσωτερικές. Μοιραστεί και ε, συμβαστική πρόταση στο άρθρο 17. Συνεχίζω. Ε, article 18 framework for... Άρθρο 18 πλαίσιο για την ανάπτυξη των ε, υποδομών προτεραιότητας. Άρθρο 20 στοιχεία υποδομών. Άρθρο 25 παράγραφος 1 οδή, θαλάσσιες οδοί, άρθρο 26 παράγραφος 2, ε, απαιτήσει υποδομών μεταφορών, άρθρο 45, απαιτήσει για το βασικό δίκτυο, εξακολουθεί η συζήτηση από αυτού, άρθρο 47 σημειώσεις για το βασικό δίκτυο. Άρθρο 49, ορισμός των διαδρόμων του βασικού δικτύου. Άρθρο 50, κατάλογος των βασικών διαδρόμων. Άρθρο 51, συντονισμός των εσωτερικών διαδρόμων. Άρθρο 54, παράγραφος 1, καταγραφή των υποχρεώσεων των κρατών μελών. Σήμερα στείλαμε στα μέλη, στους συναδέλφους, συμβιβαστικές τροπολογίες στα άρθρα 13, στο άρθρο 17, στο άρθρο 45 και σε μία σειρά από recitals 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 27, 31. Αυτά θα έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε σήμερα αλλά και σε επόμενες συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές αλλά και διμερώς ή όποιους συναδέλφους ενδιαφέρονται. Στις περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες υπάρχει μια καλή βάση, αυτό έχει προκύψει, για περαιτέρω συζήτηση και πιστεύω για σύγκληση απόψεων με τους σκιώδεις ηγητές. Τα πιο ακαθόδη ζητήματα αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή το άρθρο 13, ε, για το Comprehensive και το άρθρο 45 για το Core Network, καθώς και το άρθρο 17 που αφορά στις πλωτές μεταφορές. Αυτά είναι τα πιο ε, δύσκολα έως τώρα και τα πιο ακαθόδη ζητήματα. <coughs> τώρα, Όσον αφορά στα θεμελιώδη στοιχεία της πρώτης του κανονισμού, όπως είναι τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, οι αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία, παρατηρώ για μία ακόμα φορά ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων κινήθηκε περισσότερο με προτεραιότητες, θα έλεγα, εθνικού χαρακτήρα. Όσον αφορά ε, τις δικές μας ε, αντιδράσεις αυτά. Εμείς στηρούμε τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Προσπαθούμε να λάβουμε όσες περισσότερες ανησυχίες που έχουν καταθεί από τους συναδέλφους υπόψη μας, χωρίς όμως, και θέλω να τονίσω αυτό, να χαθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του νέου κανονισμού. Η αναζήτηση αυτής της ισορροπίας είναι και η δική μας δύσκολη θέση. Γιατί καλούμαστε και αναγκαζόμαστε να απορρίψουμε μια σειρά τροπολογιών από όλο το φάσμα των πολιτικών ομάδων, και το τονίζω αυτό, ή να δεχτούμε ορισμένες εξαιρέσεις, στη βάση όμως αυστηρών κριτηρίων και περιορισμένου χαρακτήρα. Ε, εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω ότι ε, θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση ώστε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα ε, προς την κατεύθυνση του τελικού συμβιβασμού και ενός πολύ καλύτερου και ε, ενός πολύ καλύτερου νομικού κειμένου που θα μας βοηθήσει να κάνουμε και τους κατάλληλους χειρισμούς όταν θα έρθει η στιγμή και, στην, και στον τρίλογο με το ε, Συμβούλιο. Αυτά από πλευρά μου ήταν η γενική εικόνα το που βρισκόμαστε. Ο συνάδελφος κύριος Ιωτούγκ ε, θα εμβαθύνει περισσότερο ε, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τις δικές σας παρεμβάσεις που περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ε, να σας πω ότι ο κύριος Κουμουτσάκος ε, σας παρουσίασε πού βρίσκεται η πρόοδος αυτού του θέματος. Κατά τη διάρκεια των περασμένων εβδομάδων κάναμε πολλές προσπάθειες με τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις. Όπως ήδη ακούσατε, έχουμε βρει συμβιβαστικές για τρία άρθρα, αλλά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σταθώ σε ένα πολύ, στα πιο σημαντικά άρθρα όπου μπορέσαμε να βρούμε συμβιβαστικέ. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για να διευκρινιστούν καλύτερα τα πράγματα. Καταρχήν, οι στόχοι. Άρθρα 4 και 10. Έχουμε δεχθεί μια δομή εδώ με ορισμένους στόχους, υπέρτερους στόχους όπως ε, φιλικότητα στο χρήστη και ούτω καθεξής. Αυτά τα άρθρα έχουν συγκεντρώσει πολλές τροπολογίες και γι' αυτό εμείς τη συγχωνεύσαμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες όπως εξήγησε ο κ. Κουμουτσάκος και αυτές όπως επίσης εξήγησε, έχουν τύχει συμφωνίας. Άλλες συμβαστικές προτάσεις για άρθρα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του, των σιδηροδρομικών, της κυκλοφορίας με σιδηροδρόμους δηλαδή, έχουμε πάλι για τα 14 και 15 και εκεί έχουμε ε, πολλές τροπολογίες πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε να, με τις διατυπώσεις που θα επιλέξουμε να είμαστε και συνεπείς και συνεκτική και με την ε, διευκόνηση Συνδέοντα στην Ευρώπη αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ώστε να ληφθούν υπόψη επαρκώ τα λεγόμενα μεμονωμένα δίκτυα όπου για ορισμένους συναδέλφους μας αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά και θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα είδος fine tuning για να παρουσιαστούν πιο ανάγλυφα, πιο λεπτομερώς αυτά τα ε, απομενωμένα δίκτυα ώστε όλοι να εννοούν το ίδιο πράγμα με τον όρο αυτό γιατί τώρα υπάρχουν διαφορές ερμηνείας τις βασικές πάντως ε, έννοιες τις λαμβάνουμε εδώ υπόψη και εν τέλει αγαπητοί συνάδελφοι με πολλή προσπάθεια και με μεγάλη ταχύτητα μάλιστα ήρθαμε κυρίως στο άρθρο 17 για την εσωτερική ναυσιπλογία. και εδώ νομίζω πετύχαμε έναν καλό συμβιβασμό προσπαθήσαμε με την διατύπωση που επιλέξαμε να μην προκαλέσουμε νέες απαιτήσει, νέα δηλαδή νομοθεσία που ενδεχομένως να μην συμβαδίζει με την υφιστάμενη. Γι' αυτό και παραπέμψαμε σε συγκεκριμένες ήδη υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες και έχουμε λάβει τις ε, διατυπώσεις αυτές, τις έχουμε θετήσει διατυπώσεις αυτές δηλαδή αυτούσιες. Όπως θα έχετε διαβάσει ίσως στην συμβαστική δήλωση έχουμε και αυτό το joint, joint statement για την ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Αυτό έγινε με την υποστήριξη των συντονιστών μας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες του Δούναβη και τις τρεις επιτροπές του Δούναβη. Και νομίζω ότι η βάση αυτή είναι κατάλληλη για να βασιστούμε, διότι όπως σας είπα γίνεται και δεκτή από όλους. Εξέτασα ιδίω τις τροπολογίες των συναδέλφων μου που αναφέρεται στο ε, Good Navigation Status, γιατί είναι σημαντικό αυτό για μένα και προσπαθήσαμε να το περιλάβουμε στον συμβιβασμό και με παραπομπή στην συμφωνία AGN, όπως έχει συμφωνηθεί και με τους συναρμόδιους υπουργούς των χώρων, 17, άρθρο 17.3. Και εκεί παραπέμπουμε σε εφιστάμενους ήδη ορισμούς για να μην υπάρξει κίνδυνος να σημειωθούν κάποιες ε, ασυνέπειες. Αυτά είναι τα πιο κρίσιμα άρθρα σε μια πρώτη τοποθέτηση και οι συμβαστικές προτάσεις που είχαμε υποσχεθεί και που τις υποβάλλουμε σήμερα. Αναμένουμε βεβαίω μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις αλλά και άλλες προτάσεις για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Αύριο θα έχουμε την επόμενη συνάντηση των σκιωδών και στις 12 Δεκεμβρίου θα ξανασυναντηθούμε με του Σάντο για να συζητήσουμε την τελική μορφή του κειμένου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε εγκαίρως μέχρι 18-12 να έχουμε φτάσει σε μια τόσο καλή μορφή του εγγράφου που να μπορεί να βρει σύμφωνους πολλές και πολλούς από τους συναδέλφους μας. Μέχρι τότε ωστόσο είμαστε στη διάθεσή σας για συζήτηση και αναμένουμε την επικοδομητική σας ε, υποστήριξη. Σας ευχαριστώ. Έχω τον κύριο Μπιλμπάου, τον κύριο Κράμερ, Αλκατράουι, Μπέρκ, Μπραντμπον, Αγιάλα, Ντεμπάκ, Σεβεράμα, Ντεγκράντες, άλλος στον κατάλογό μου γιατί όσο πιο πολύ μακραίνει ο κατάλογος τόσο λιγοστεύει ο χρόνος. Mr. Kuhn, Mr. Udias, and Mr. Benyon. So you have about 10 seconds each. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's 14 speakers. Κατέσσερις ομιλητές έχω. Δύο λεπτά έκαστος. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα δύο λεπτά που μου δίνετε. Όπως είπαν και οι συγγητές, έχουμε κάνει πολλή δουλειά και η ομάδα μας στήριξε τις συμφωνίες πλήρως. Νομίζω ότι δέχτηκαν και συγκητές συμβασμούς, οπότε υποστηρίζουμε την μεθοδολογία που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνούμε να διατηρήσουμε τις προθεσμίες και επιπλέον ενισχύσαμε και τις έννοιες της ε, προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας, ε, το θέμα του cross-border, την ε, παρουσία και την ανάγκη ύπαρξης μιας διακυβέρνησης όπου να συμμετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και την ανάγκη να υπάρχει συντονισμός σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να σας πω ότι αν μη τι άλλο οι συμβασμοί που είδαμε μέχρι τώρα και από τις συζητήσει που κάναμε μέχρι τώρα η ομάδα μας κατάφερε να συμφωνήσει. Υπάρχουν σήμερα οι συμβασμοί που πρέπει βέβαια να τους κοιτάξουμε με λεπτομέρειες, αλλά γενικά η στάση μας είναι θετική. Ναι στη μεθοδολογία, ναι στις προθεσμίες και η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να εγκριθεί στις προθεσμίες που αναφέρονται χωρίς καθυστερήσεις. Συμφωνώ και με τις πλωτές οδούς. Θα ήθελα βέβαια να ξέρω για τον κατάλογο, αν υπάρχει κάποια αξιολόγηση μέχρι τώρα. Από πλευρά μου, τίποτα άλλο και έχω σεβαστεί και τα δύο λεπτά που μου δώσατε. Ευχαριστούμε ο κύριος Κράμερ. Και εγώ ευχαριστώ τους δύο συντονιστές, το συντονιστές γενικά, το πρόβλημα που έχουμε εμεί είναι ότι πρέπει να γίνει και μια αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων. Οι τιμές δεν είναι ορθές. Ούτως ή άλλως δηλαδή τελικά θα προκληθεί το διπλό κόστος και ο διπλός χρόνος θα χρειαστεί. Δεν έχουμε όμως χρόνο. Δεν προλαβαίνουμε να προστατεύσουμε το κλίμα για τα cross-border, συμφωνώ. Χρειαζόμαστε όμως τον ίδιο ορισμό. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικά, διαφορετικούς ορισμούς και διαφορετικά κριτήρια στα διάφορους ε, φαγγέλους. Για τα missing links, πράγματι εδώ πρέπει προτεραιότητα να πάρει ο σιδηρόδρομος. Αλλά πιο πολύ χρειάζεται συντήρηση και εδώ υπάρχει μια διαφορά στη γερμανική ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στη μετάφραση και η οποία θεωρώ ότι δεν είναι σωστή. Ακούσαμε και για τα καλαπέ, είπατε ότι ρόλος, ο, το χρήμα δεν παίζει ρόλο, ότι θέλουν να είναι πλωτοί οι ποταμοί ολόκληρο το έτος και τι γίνεται, κάποιες μέρες δεν είναι, γύρω στις 60-65 μέρες το χρόνο δεν είναι πλωτοί οι ποταμοί και μέχρι ότου γίνει πλωτός ο Δούναβης αλλά δεν θα προλάβουμε να τα δούμε εμεί όλα αυτά τα πράγματα, ούτε καν τα παιδιά μα νομίζω, γιατί είναι πολύ δαπανηρέ οι επενδύσει αυτέ. Σε αυτά πρέπει να συμβάλλει ο σιδηρόδρομο. Αυτό που λείπει εδώ είναι ότι δεν περιλαμβάνεται ο στόχος της μείωση του 20% μέχρι το 2020, ενώ στο ΣΕΦ είναι μέσα. Τα εθνικά κριτήρια και εθνικοί εγωισμοί δηλαδή, φαίνεται, φαίνονται αυτά και από τις χιλιάδες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Είναι σαφές ότι τέτοια πράγματα δεν έχουν χώρο, σε δεν έχουν τόπο μάλλον σε ένα ενιαίο ε, ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Τέλος, δεν βλέπω ποδηλατόδρομους. Είναι όμως μέσα στον, ε, στο λευκό βιβλίο. Και αυτά είναι και αυτά διάδρομοι. Είναι 70 χιλιόμετρα. Τα ακούσαμε και άλλη φορά. Η δεύτερη γέφυρα μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας είναι σημαντική και για τον Δούναβη και για τις ε, παραπλήσεις περιοχές. Πρέπει να μπει μέσα. Πρέπει να σκεφτούμε συντονισμένα. Για το Σαβαρή το σκεφτήκαμε τελευταία στιγμή και πίστηκε ότι είναι σημαντικό και σωστό. Παρακαλώ να περιληφθούν λοιπόν και οι ευρωποδηλατόδρομοι. Ορισμένε χώρες μέλη με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να προσπαθήσω να τα περάσω. Δεν είναι λοιπόν θέμα μοναχά των πράσινων. Okay. Uh, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για τη μεθοδολογία που ακολούθησαν, για την υπομονή τους έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό. που συνδυάζεται βέβαια στο τόχο μας να μείνουμε στη μεθοδολογία που έχουμε αποφασίσει από τη μια και από την άλλη μεριά το περιθώριο που παραμένει να είναι όσο γίνεται πιο ευρύ, η ερμηνεία δηλαδή να μπορεί να είναι όσο γίνεται πιο ευρύ έτσι ώστε οι συνάδελφοι με επικοδομητικές προτάσεις να μπορέσουν να βοηθήσουν. Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πολύ. Βέβαια καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είναι κανεί 1000% ικανοποιημένο, πολύ να είναι απογοτευμένοι με τα πράγματα που έχουμε τώρα μπροστά μας, αλλά εγώ πιστεύω ότι αποτελεί ένα καλό συμβαστικό πακέτο. Παραμένουν κάποια θέματα που θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες δίχως άλλο για τις εσωτερικές, ε, την εσωτερική ναυσιπλοεία. Τα είπαν και οι συγητές ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανησυχίες του κλάδου και συγχρόνως να λάβουμε υπόψη μας και τα περιβαλλοντικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις επόμενες εβδομάδες και στις 18 Δεκεμβρίου που θα ψηφίσουμε πιστεύω ότι τελικά θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα ως ε, κοινοβούλιο και θα έχουμε κάνει ένα νέο βήμα προς ε, ένα αξιόλογο στοιχείο των ευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά ο κύριος ε, Πίρκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στους δύο σχητές για την συνεργασία και το πνεύμα προς συνεργασία. Έρχομαι όμως στον συμβασμό για το άρθρο 5 όπου λέει ότι στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των έργων θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το στοιχείο αποδοχής από μέρους των πολιτών και στον σχεδιασμό ιδίω να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα οι τοπικές ιδιαιτερότητες για την χάραξη των ε, ε, διαδρομών. Εφόσον πράγματι οι χώρες μέλη οφείλουν να το λάβουν αυτό υπόψη, θα πρέπει τότε να είναι δυνατόν να γίνουν και εναλλακτικέ προτάσεις, ε, με λεπτομέρεια δηλαδή. Εκεί θα πρέπει να αναμένεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία που να δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία ιδιαίτερα για ορεινές περιφέρειες ή περιφέρειες με ιδιαίτερο φυσικό κάλος ή τουριστικό ενδιαφέρον. Υπάρχει λοιπόν η τροπολογία 75 νομίζουμε είπε ο που θα ήθελα το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος της που λέει ότι οι χώρες μέλη εφόσον είναι απαραίτητο προτείνουν εναλλακτικές διαδρομές ή εναλλακτικά μέτρα. Αυτό αποτελεί συνέπεια από το πρώτο. Πρόκειται για μια διευκρίνηση και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα η, ο σκοπός δηλαδή της αποδοχής από τους ενδιαφερόμενους και να μην υπάρξουν τόσες πολλές αντιδράσεις από τους ε, ενδιαφερόμενους πολίτες. Παρακαλώ να περιληφθεί λοιπόν και το δεύτερο μέρος αυτής της τροπολογίας.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 αναρωτήθηκε πώς θα ευθυγραμμίζεται το κείμενο στο πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων με τις τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας. Το Connecting Europe είναι ένα στοιχείο κλειδί. Και εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες και αντιλαμβάνομαι τα σχόλια, αλλά δεν βλέπω συγκεκριμένη σύνδεση Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω για να δούμε τεχνικά πώς θα πετύχουμε, δεδομένου μάλιστα, Πρόεδρε, ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερες περικοπές στον προπολογισμό. Τα ακούσαμε και από, το... από τις συζητήσεις που έγινε για τον προπολογισμό με τον κύριο Φανεροπάου την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, αν μη τι άλλο, να φροντίσουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τέλο πάντων η πτυχή αυτή, να είναι ρεαλιστική. Τώρα για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες αυτές καθ' αυτές. Εντάξει, αλλά υπάρχει μια τάση. Ξέρετε εξάλλου, Πρόεδρε, ότι ήμουν εισηγητή στο προηγούμενο πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων. Ε, λοιπόν, πολλέ από τι συμβαστικέ προτάσει που βλέπω εγώ είναι σαν ε, πάλι δέντρο. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην ανακατεύουμε όλες τις ιδέες αλλά να έχουμε έναν ευρύ ορισμό του τι θέλουμε να πετύχουμε με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δηλαδή, με δύο λόγια, πρόεδρε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι είναι εφικτό και τι όχι, κατά πόσο μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά τα προγράμματα. Και βέβαια, όπως είπα και πριν, να λάβουμε υπόψη μας τους οικονομικούς περιορισμούς, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Άκουσα σχόλια για να πετύχουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτή η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης είναι κάτι που το έχουμε κάνει καραμέλα. Προσοχή όμως, τι ακριβώς εννοούμε με αυτό. Μην βάζουμε προσδοκίες που τελικά δεν ισχύουν. Πολλές φορές είναι περισσότερο διαφήμιση παρά πραγματικά προστιθέμενη αξία. Το άλλο που θέλω να πω, Πρόεδρε, και πάλι το λέω από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι βλέπω πολλές συμβαστικές τροπολογίες για τα παραρθήματα. Λέω προσοχή. Ώρες και ώρες έχω περάσει τα τελευταία 7-8 χρόνια για να οργανώνω τέτοια πράγματα. Προσοχή λοιπόν, γιατί κάθε φορά που προσπαθείτε να τροποποιήσετε ένα παράρτημα, τελικά αντικαθιστάτε ένα παράρτημα από ένα άλλο. μια που υπάρχουν επιπλέον ε, προτεραιότητες. Και το θυμάμαι, να... το έχω πάθει και εγώ αυτό με το προηγούμενο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα έλεγα πολύ προσοχή κάθε φορά που θέλουμε να τροποποιήσουμε ουσιαστικά τα παραρτήματα ή να προσθέσουμε κάτι. Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό δηλαδή, γι' αυτό το λέω, όχι τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόντ. Ήμουνα γενναιόδωρος μαζί σας. Χρωστά στο κύριε Μπιλμπά λεπτό τότε. Ο κύριος Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τα όσα μας είπαν και για τη δουλειά που κάνανε στην υπόθεση αυτή. Ως σκιώδης ε, εισηγητής θέλω να σας πω πως πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ μας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Είναι κάτι που το συζητάμε και στα πλαίσια του Connecting Europe αλλά πρέπει να είμαστε πράγματι ρεαλιστές στην ε, πρότασή μας. Δεν θα αναφερθώ σε όλους τους συμβασμούς, αλλά σε μία τροπολογία. Για τον ε, κατάλογο με τους εσωτερικούς ε, λιμένες. Υπάρχει μια θετική προσέγγιση, αλλά εδώ πέρα πρόκειται για έναν κατάλογο, ο οποίος θα πρέπει να είναι σαφής, ενώ τώρα δεν είναι αρκετά σαφής πιστεύουμε. Το Συμβούλιο επίσης έχει ένα κατάλογο, η Επιτροπή συμφωνεί, ίσως θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να μπει σε μια ξεχωριστή συμβαστική τροπολογία ο κατάλογος αυτός. Πάντως υπάρχουν και καλοί συμβιβασμοί για τα άρθρα 17 για παράγραφος 3α Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το περιβάλλον, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι μερικές φορές όλες αυτές οι παραβολητικές μελέτες δεν ε, θα ισχύουν απαραίτητα και στο μέλλον. Μια τελευταία παρατήρησή μου έχει να κάνει με κάτι που είπαν και άλλοι. Υπάρχει μια τάση να γεμίσουμε το κείμενο με εξαιρέσεις, όχι μόνο τεχνικού χαρακτήρα, αλλά για να λάβουμε υπόψη μας εθνικές ιδιαιτερότητες. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να περιοριστούμε όσο γίνεται και να μην βάλουμε τα εθνικά συμφέροντα να έχουν το πάνω χέρι απέναντι στα ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπάκερ. Ένα λεπτό και 59 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Φοβερή επίδοση. Η κυρία Γιάλα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές για τη δουλειά τους, την τόσο λεπτομερή και δελεχή όσον αφορά τις συμβαστικές προτάσεις. Ιδιαίτερα ευχαριστώ για την πρόταση που έχει γίνει όσον αφορά τη ρήτρα αναθεώρησης. Στο άρθρο 57 δηλαδή, όπου υπάρχει μια πρώτη βάση για συμβασμό σε σχέση με τα κατά προγράμματα τα οποία για διαφορετικούς λόγους δεν έχουν μπει ακόμα στην αναθεώρηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και κάτι. Γιατί δεν λάβατε υπόψη σας τον ορισμό της διαλειτουργικότητας. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον αυτό. Γιατί δεν βάλατε τη διαλειτουργικότητα λοιπόν. Και κάτι άλλο τώρα όσον αφορά τα παραρτήματα. Ελπίζω μετά από όσα καταφέραμε να βάλουμε οι Σουηδοί για παράδειγμα και άλλα που ξεχάσαμε, ελπίζω ότι και με τον Νότο θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε κάποιες πτυχές. Το οροδρόμο του Ντεβίγου για παράδειγμα ή άλλα. Τώρα όλος ιδιαίτερος θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με το παράρτημα 1, τη συμβαστική πρόταση εκεί για το 533, βλέπω ότι εκεί αναφέρεται ο δρόμος Αρούς Χιστάλ και θέλω να ρωτήσω. Εγώ νόμιζα ότι δεν αποτελούσε μέρος της μεθοδολογίας να συμπεριλάβουμε οδούς ή τμήματα δρόμων. Και αυτό θα ήθελα λοιπόν να μου το εξηγήσετε γιατί το κάνατε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και άλλοι περιμένουμε και θα θέλαμε να βάλουμε μέσα ε, οδικές αρτηρίες. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε γιατί. Τέλος. Οι τροπολογίες, τις συμβαστικές, κάποιες έχουν σελίδα, κάποιες δεν έχουν. Ε, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποια είναι η διαφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λίχτεμπεργκερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Γενικά πρώτα, θυμίζω ότι πέρσι είχαμε την έκθεση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που είχα συντάξει εγώ ίδια και είχε εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Από τις προθέσεις που είχαν περιληφθεί σε αυτήν την έκθεση τότε, δηλαδή μια συγκέντρωση στα πιο σημαντικά, μια βελτίωση των διασυνδέσεων των κομβικών σημείων μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, δυστυχώς δεν παρέμειναν πολλά, δεν διατηρήθηκαν πολλά. Παραδείγματα. Ήδη τότε και τώρα πάλι στο σχέδιο είχαμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχουν ε, οδοί που να συνδέουν με τις μεγάλες αρτηρίες. Εφόσον αυτά θα μας φάνε ούτως ή άλλως τα δύο τρίτα των ε, κονδυλίων που θα μας μείνουν μετά για τα διευρωπαϊκά έργα. Βλέπω εγώ σε γερμανική εφημερίδα εδώ ότι για την ε, διαδρομή Μόναχο-Ζυρίχη η ηλεκτροδότηση θα γίνει το 2020. Διερωτώ με, τι μιλούμε, τι συζητούμε εδώ. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση σε όλους και όλους ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε μην πάμε να φτιάχνουμε κάστρα στην άμμο. Είναι απαραίτητες οι διαδρομές αυτές που οδηγούν στις αρτηρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. εξέτασα το θέμα με τις αρχές της Ελβετίας και της Ιταλίας. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν τις ε, απαραίτητες διασυνδέσεις με τον σιδηρόδρομο, με τις αρτηρίες του σιδηρόδρομου. Δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνομαι, αλλά εδώ οφείλω να το πράξω, διότι αλλιώ όντω φτιάχνουμε καθεδρικού στην άμμο, στην έρημο. Και μια φράση ακόμα για το Ευρωβελό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τουριστική σημασία. Το ίδιο τουλάχιστον όπω το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Γιατί λοιπόν το ένα είναι μέσα και το άλλο έξω. Σαβάμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ Θέλω να απηχήσω τόσο είπε ο κ. Χέρτζοξ και εγωγικές του Πατρίζη. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφεί για το τι συζητάμε. Μιλάμε για τεχνικές προδιαγραφέ, αλλά αν υπό το άρθρο 13 μπορεί να είναι αυτονόητο τι σημαίνουν μεμονωμένα, απομονωμένα δίκτυα, υπό το άρθρο 45 Εκτός και αν έχουμε τα πάντα στο ε, σκέψη, στην οποία αναφέρεται το κείμενο, ανησυχώ πως η παράγραφος 2α για τις σιδηροδρομικές υποδομές, εκτός από τα απομονωμένα δίκτυα, εκεί πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση για το τι ακριβώς σημαίνει εκεί αυτή η φράση, να ξέρουμε δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε. Ευχαριστώ. Εγώ μπορείτε να δώσετε ένα λεπτό μου στην ε, κυρία Μπιλμπάου. Η ε, κυρία Μπιλμπάου θα έχει τόσο πολύ χρόνο στο τέλος. Ο κύριος Δεγκράντες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πω σύντομα. Καταρχήν, συμφωνώ από το Α μέχρι το Ω με την παρέμβαση του Ε, με, τις, ε, συντονιστές, με τους ε, εισηγητές με συγχωρείτε, αλλά διαφωνώ με την κυρία Μπιλμπάου και κυρίως με τον κύριο Κουμουτσάκο που είπε ότι πρέπει να είμαστε όντως ευέλικτοι και, το, ευέλικτοι και το έπραξε αυτό ο κύριος Κουμουτσάκος και έπειτα παρά τη δουλειά που έχετε κάνει και σας ευχαριστώ και εκτιμώ το η δουλειά που κάνατε δεν μπορούμε ακόμα να πούμε πως είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Δεν είμαστε ακόμα ευχαριστημένοι σε αυτό το στάδιο. κυρία Σανάλοβα, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θέλω να αναφέρω τρεις παρατηρήσεις σε τρεις τροπολογίες. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για τη δουλειά τους, για τις συμβιβαστικέ. Επίσης, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω για το άρθρο 3 ε, όπου πραγματικά αφηνίζεται τι υποτίθεται ότι είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Έπειτα να αναφέρω και την συμβαστική του άρθρου 17, όπου εκτιμώ την προσπάθεια που κατέβαλαν οι συνεισηγητές, αλλά νομίζω πως πρέπει να είμαστε συνεπείς και να μείνουμε στην ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και να μην εκτεθούμε σε υποκειμενικές αξιολογήσεις. Αυτό ήταν ιδιαίτερο ατυχές. Και τέλος για το άρθρο 57 και τη σχετική συμβιβαστική και εκεί ε, φαντάζομαι πως θα χρειαστεί να κάνω μια πιο αποδεκτή διατύπωση ώστε να ληφθούν υπόψη και τα διασυνοριακά προγράμματα που βρίσκονταν στο στην αρχική απόφαση ε, του 2010 για τα TEN-T. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συνεισηγητές που εργάστηκαν με ακριβή τρόπο και έχουν λάβει αποφάσεις οι οποίες είναι και εύλογες. Τα τεν έχουν μια νέα ποιότητα απέναντι στην προηγούμενη συστηματική κατάταξη που προηγουμένως είχαμε ένα διαφορετικό, μια διαφορετική δόμηση και τώρα έχουμε δίκτυα με κομβικά σημεία που για αυτά, για αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουν λεχθεί τα σχετικά με τα προηγούμενα τώρα. Εάν θέλω να φτιάξω μια αρτηρία, πρέπει πρώτα να εξαλείψω τα μεγάλα εμπόδια. Πρέπει να ξεπεραστούν από βορρά προς νότον, για παράδειγμα, τα μεγάλα ποτάμια, τα ε, βουνά, τούνελ στον άξονα από δυσμόν προς Ανατολάς, αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν και υπερβολικές επιβαρύνσεις. Έχουμε τα επόμενα 10 χρόνια να περιμένουμε 20% αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών. Και βέβαια και η πρόκληση θορύβου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό χαίρομαι που έγινε ένα από τα κριτήρια και δεν μιλούμε μόνο για, για Genoa Rotterdam, αλλά μιλάμε και για ανατολικά προσδυτικά πλέον καθώς επίσης και για τον άξονα προς τη Σκανδιναβία, είτε περνάμε από Αμβούργο, είτε από Ρόστοκ, είτε από Γκτάνσκ στην Πολωνία, όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Και για το περίφημο Motorways of the Sea, επίσης χαίρομαι και ευχαριστώ που το περιλάβατε, χρειαζόμαστε ένα αποδοτικό δίκτυο. Μας λείπουν βέβαια κάμποσα κονδύλια. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη ότι θα προχωρήσουμε και στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Βλέπω τον Μάικλ και την κυρία. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ούτζιας. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές και τους Κεώδης μεταξύ και αυτών και την κυρία Μπιλμπάου για την ε, αφοσίωσή τους. Νομίζω πως η πρόταση που προέκυψε είναι ισορροπημένη με την ένταξη των συμβατών συμβιβαστικών με βάση τις μεθοδολογικές εντολές που τους δόθηκαν. Φυσικά ο καθένας από εμά θα, ήθελε να βάλει κάθε περιφέρεια, κάθε υποδομή, αλλά με, τότε θα ήταν ένα δίκτυο εξαιρετικά ευρύ Όλοι όμως εδώ αντικατοπτρίζουμε γενικά συμφέροντα και το κοινό συμφέρον. Πάντως η πρόταση είναι σημαντική για ένα σύνολο. Δείχνει πώς μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μου για την αποδοχή των ε, τροπολογιών που υποδεικνύουν ένα σύνολο, ένα σύστημα συνολικό. Και επίσης έχουμε και μια βελτίωση στο κομμάτι εκείνο της πρότασης όπου συμπεριλαμβάνονται ε, το σύστημα με τα μεγάλα νησιά, η Κρήτη, η Σαρδινία, ε, με την συμπερίληψη του Ηρακλείου και του Κάλιαρη και του Λιμένα και του Αερολιμένα. Και ε, γι' αυτό θα σας πω ότι είμαι ικανοποιημένο και στηρίζω την πρόταση. Ευχαριστούμε κύριε Ούτζες. Κύριε Ζεβέντκεν, ευχαριστώ. Εγώ δεν θα μιλήσω για πολλή ώρα. Αυτό το περιθώριο ασφαλείας που λέτε 10 μέτρα ασφαλείας, δεν, δεν κατάλαβα ακριβώς από πώς που είναι αυτά τα 10 μέτρα, εν πάση περιπτώσει μάλλον θα ξέρετε κάτι. Υπάρχουν όμως ε, λειτουργικές δυσκολίες γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα 10 μέτρα. Αν μπορούσατε να, να με ενημερώσετε. Το δεύτερο σημείο είναι για το ανάπτυξη του RTMS. Είμαι υπέρ της ανάπτυξης του. Τώρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν εθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη του RTMS, αλλά από τη στιγμή που αυτά τα προγράμματα είναι λογικά, εντάξει. Αλλά το να κάνει κανείς ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί μετά να υλοποιήσει, δεν έχει νόημα. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα όμως, θα πρέπει να αλλάξει ώστε να ταιριάζει στην αρχή αυτών όσων προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή εδώ κάποια ευελιξία. Και τρίτον, έχω πρόβλημα με το κείμενο όσον αφορά το άρθρο 49 που λέει ευθυγράμμιση των ε, διαδρόμων των σιδηροδρομικών θα αλλάξει ώστε να αντιστοιχεί στην ευθυγράμμιση των οδικών βασικών διαδρόμων. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Αν ο διάδρομός σου για σιδηροδρομικές μεταφορές ε, προϊόντων φτάνει και αφήνει μια γραμμή περίπου 10 χιλιόμετρα μάκρους, τι σημαίνει ότι αυτό πρέπει να κατασκευαστεί κάπου αλλού, σε κάποιο διαφορετικό μέρος. Αν αυτό το ερμηνεύσει δηλαδή κανείς στην κυριολεξία, μπορεί να υπάρξουν πολλές ε, ε, αχρίαστες δαπάνες, περιττές δαπάνες. Όπως τώρα είναι διατυπωμένο, φαίνεται σαν να ζητά κάποια μάλλον ανόητη ευθυγράμμιση, ε, και όπου αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί όμως να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Μπορούμε κάπως να το διατυπώσουμε διαφορετικά ώστε να είναι λογική η πρόταση. Ευχαριστώ για να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Είναι μια ερώτηση σειροδρομικού τύπου και θα πρέπει να ξέρω την απάντηση. Είναι η απόσταση ανάμεσα στο τέλος του τρένου και στο τέλος της ε, προβλήτας. Ε, δέκα μέτρα απόσταση ε, από το σταθμευμένο τελευταίο βαγόνι και το επόμενο, έτσι ώστε να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στα τρένα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τους ε, συνεισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές για την προσπάθειά τους. Υπάρχουν κάποια σε ακόμα συνεδριάσεις μέχρι που να ψηφίσουμε, ώστε να, έχουμε, να φτιάξουμε ένα κατάλογο ψηφοφορίας ε, που να μπορούμε να το διαχειριστούμε, γιατί ο δικό μου εφιάλτης αυτό είναι. Και επανέρχεται στα όσα είπα στην αρχή. Ο κύριο Μπράτμπορν είπε και σωστά, και η κυρία Λίχτεμπεργκερ το έθιξε αυτό σωστά. Ε, γιατί θυμάμαι το την πρώτη ψηφοφορία για τα TNT στις αρχές του 90. Ήταν ένα ευχολόγιο για τα Χριστούγεννα, για τον Φίλιπ, για, τον, για την Ήβα. Ναι, εδώ κινδυνεύουμε. Κινδυνεύαμε να έχουμε ένα ευχολόγιο. Ναι, κινδυνεύαμε και αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Και χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να το καταφέρουμε αυτό. Είπαμε, φτιάξαμε τη μεθοδολογία, ξέρουμε ποια είναι η μεθοδολογία με την οποία δουλεύουμε. Αν εντάσσεται στη μεθοδολογία, τότε οι εισηγητέ ήταν αρκετά βοηθητικοί και το έχουν συμπεριλάβει στην τροπολο... στην συμβιβαστικές. Αν όχι, κατά τη γνώμη μου, σωστά δεν θα πρέπει να είναι μέσα. Και αν δηλαδή περάσει η συμβιβαστική θα πρέπει να καταπέσουν τα υπόλοιπα. Κυρία Μπιλμπάου, θα σας δώσω ένα άλλο ένα λεπτό, γιατί ξέχασα πως ήσασταν σκιώδη συγκέτρια. Γι' αυτό σας δίνω ένα παραπάνω λεπτό, κυρία Μπιλμπάου. Σας υπόσχομαι, Πρόεδρε, ότι το σημαντικό δεν είναι πόσο χρόνο μιλάμε, αλλά το τι λέμε, ακόμα και αν μιλάμε λιγότερο. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω είναι ότι άκουσα τον κύριο Λουίς Γκράντης, και εγώ συμφωνώ με τους ε, εισηγητές μας και το είδα αυτό στις τέσσερις συναντήσεις που κάναμε ότι η μεθοδολογία, η προστιθέμενη αξία, η νέα διακυβέρνηση, η υποχρέωση τέλος πάντων η προσπάθεια για να τηρήσουμε τις προθεσμίες για να κάνουμε μια σοβαρή πρόταση, όλος ανέφερα και πριν όταν πήρα το λόγο, συνάδουν απόλυτα με το έργο μας και με τις συμβατικές προτάσεις τις οποίες καταλήξαμε με τους εισηγητές. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Καλώς. Κύριε Δεγράντες, με που αναφέρθηκε το όνομά σας, έχετε το δικαίωμα να απαντήσετε αν θέλετε. Όχι. Καλώς. Είναι. Α. Ναι, ναι, κυρία Μπιλμπάο, δεν πρόκειται να τσακωθώ τώρα μαζί της. Το μόνο που θα πω είναι ότι ότι θα αποδειχθεί στην πράξη το τι θα κάνουμε. Ήταν ισπανική η παροιμία που είπατε και μάλλον ε, δεν είναι σίγουρο ότι μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες. Και εγώ το ίδιο παθαίνω, λέει ο πρόεδρος. Κάθε φορά που λέω μια αγγλική παροιμία είναι δύσκολη μετάφραση. 30 δευτερόλεπτα εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ε, εισηγητές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για να συνεχίσουμε την τεχνική δουλειά που θα χρειαστεί στη συνέχεια μέχρι την 18η του μηνό, στην ψηφοφορία δηλαδή. Καλώς. Οι εισηγητές τώρα. Ο κύριος Κουμτσάκος πρώτα για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ε, το εξής, ότι οι συμβαστικές προτάσεις είναι ακριβώς αυτό το οποίο δηλώνει η λέξη. Συμβιβασμοί. Δεν παρέχουν 100% ικανοποίηση σε κανέναν. Αλλιώς δεν θα τους λέγαμε συμβασμούς. Έτσι έχουμε προχωρήσει σε αυτή την Επιτροπή για όλα τα θέματα που έχουμε συζητήσει και αποφασίσει. Αυτό θα ισχύσει και σε αυτό το νομοθετικό κείμενο. Οι συμβιβασμοί λαμβάνουν υπόψη και κάναμε ό,τι μπορούμε για να λάβουμε υπόψη τις βασικές ανησυχίες, τις βασικές προτεραιότητες που όμως είναι σύμφωνες με τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι 100% ικανοποιημένος, τότε δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας εμείς, οι εισηγητές. όσον αφορά τους ποδηλατόδρομους. Ε, σίγουρα δεν είναι θέμα του κόμματος των Πρασίνων. Το ποδήλατο είναι ένα όλο και πιο λαοφιλές ε, μέσο και οπωσδήποτε δεν ανήκει σε καμία πολιτική ομάδα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Βέβαια, το ποδήλατο είναι ένας κατά βάση τρόπος μεταφοράς που συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στην άθληση και δευτερευόντως στη μεταφορά. Και τουλάχιστον εκεί μπορούμε νομίζω όλοι να συμφωνήσουμε. Σας καλώ λοιπόν όλους τους Γερμανούς επισκέπτες της Κρήτης να έρθετε στο αναβαθμισμένο εξανάγκης αεροδρόμιο του, του Ηρακλείου και να κάνετε ποδήλατο στην Κρήτη. Λοιπόν, όσον αφορά ε, τα, το, όσον αφορά τα θέματα του δικτύου τώρα των ποδηλάτων, θέλω να πω το εξής. Έχουμε λάβει υπόψη μας στο δίκτυο ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η ασφάλεια με τις διασταυρώσεις με ποδηλατόδρομους. Αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αλλάξουν οι χάρτες και να συμπεριληφθεί το δίκτυο του ποδηλατόδρομου στους χάρτες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Δεν είναι γιατί αυτό είναι μια θέση μας εναντίον των ποδηλάτων, αλλά γιατί νομίζω ότι θα κινηθούμε πολύ πέραν, πολύ πέραν του σκοπού και του στόχου του κανονισμού τον οποίο συζητάμε. Άλλωστε αυτό έχει να κάνει και με την χρηματοδότηση. Όταν όλοι συμφωνούμε ότι κινδυνεύουμε να έχουμε μια ελληματική και όχι επαρκή χρηματοδότηση, νομίζω ότι είναι περίεργο την ίδια στιγμή που συμφωνούμε αυτό να προσθέτουμε ή να θέλουμε να προσθέσουμε και, άλλα και προοπτική άλλων έργων που ξέρουμε δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Υπάρχει μπροστά μα και νομίζω ότι τη συζήτηση μπορούμε να την κλείσουμε εδώ με καλή πίστη. Υπάρχει μπροστά μα νομοθετικό κείμενο που θα αφορά μόνο, μόνο τους, πολυ... Εκεί πέρα θα καταγραφούν και οι πιο φιλόδοξες και οι πιο ρεαλιστικές προτάσεις. Και ας μην ξεχνάμε ότι το 23 προβλέπεται, υπάρχει η ρήτρα αναθεώρησης των διευρωπαϊκών δικτύων. Ας δούμε ποια θα είναι η πολιτική δυναμική της εποχής, ας δούμε ποια θα είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των ε, κατευθυντηρίων γραμμών που συζητάμε σήμερα και η συζήτηση μπορεί να ξανανοίξει. Αν και εγώ πιστεύω ότι, ότι επί της αρχής στο στάδιο αυτό δεν μπορούν οι ποδηλατόδρομοι να εντάσσονται στο δίκτυο. Ε, όσον αφορά την ε, τροπολογία 275, την άκουσα με προσοχή την πρότασή σας, θα πρέπει ακριβώς να δούμε <clears throat> ποιες μικρές ε, διαφοροποίησεις πρέπει να γίνουν ώστε ε, να καλυφθεί και η δική σας ανησυχία. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι ακριβώς το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 275 ε, νομίζω ότι δεν μπορεί ακριβώς ως έχει να ενταχθεί. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα έχουμε ένα πεδίο που θα βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Συμφωνώ με τον κύριο Μπράντμπον στη βασική τη λογική. Ε, πρέπει να είμαστε αυστηροί, πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε. Έχουμε κάνει εξαντλητικές συζητήσεις σε όλα τα θέματα, με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ακόμα φτάσαμε κι εμείς οι εισηγητές να κάνουμε πίσω από τον πυρήνα των θέσεών μας. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την ευελιξία ε, στα βασικά θέματα εννοώ, στα θεμελιώδη θέματα, από εκεί και πέρα στα περιφερειακά θέματα και στις περιφερειακές ανησυχίες είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε, μια, ε, σε έναν αποδεκτό συμβασμό. Τέλος, όσον αφορά τον κατάλογο με τους βασικούς λιμένες, ε, μπορώ να πω ότι αυτός ο κατάλογος βρίσκεται στο δρόμο να ενταχθεί στο κείμενο. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω και να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι ο συμβιβασμό είναι ακριβώ αυτό το οποίο λέει, η λέξη. Συμβιβασμό. Και θα παρακαλέσω όλου του συναδέλφου σε αυτή τη λογική να κινηθούν ώστε να καταλήξουμε μαζί στο καλύτερο δυνατό κείμενο. Αν αναφέρθηκα λίγο κουραστικά στην αρχική μου εισήγηση σε, όλα τα, σε όλες τις τροπολογίες και σε όλους τους συμβασμούς είναι για να ακουστεί πόση προσπάθεια έχει γίνει και από εσάς και από εμάς. Παρακαλώ, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες στη διάθεσή μας. Ελπίζω ότι θα επιτύχουμε ένα πολύ καλό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε να προσθέσετε τίποτα κύριε Ερκούτ. Όχι, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και και τους συναδέλφους. Θα κάνω μια σύντομη σύνοψη των όσων εξηγήσατε εσείς και εσείς κύριε Πίρκερ μιλήσατε για την 275 το δεύτερο μέρος θα επανέλθουμε και θα σας εξηγήσουμε ο κύριος Ντεπάκερ μίλησε για τον κατάλογο των ε, λιμανιών εσωτερικής ναυσιπλογία. μόλις απάντησε ο κύριος Κουμουτσάκο. εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι στόχος μας είναι να υπάρξει σαφήνεια ώστε καθένας που όπως για παράδειγμα σε Ολλανδία και Βέλγιο είναι δύσκολο να αντιλαμβάνεται κανείς ποια λιμάνια εννοούνται, γι' αυτό το περιλάβαμε. Αυτό ισχύει όχι μόνο για, τα εσωτερικά, για λιμένες, αλλά και για τα αεροδρόμια και για τους τερματικούς σταθμούς σιδηροδρόμων. Πληροφορία ωστόσο και σαφήνεια πρέπει να είναι πρώτη στόχος. Η κυρία Ιάλα Σέντερ μίλησε για ένα τμήμα του δρόμου, αλλά δεν ήταν απόλυτα σαφές για μένα, ίσως ήταν και πολύ ε, γρήγορη, γρήγορος ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, αλλά αν θέλει διμερώσεις μπορούμε να ε, διευκρινίσουμε το θέμα. Μιλήσατε και για την διαλειτουργικότητα στον σιδηρόδρομο, είναι το 12, 30 και 55, αυτά τα άρθρα αναφέρονται σε αυτά. Αύριο θα ξανασυζητήσουμε πάλι με τους εσκιώδεις και νομίζω ότι θα σας ικανοποιήσει αυτό που θα συμφωνήσουμε, αν και δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει. Για τα παρατήματα, για το θέμα αυτό, στο παρατημά μας έχει μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα. Μόνο δηλαδή για αποσαφήνιση και δεν θέλει διόλου να μπει στις αρμοδιότητες της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Το λέω αυτό για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ μίλησε για τις ε, γραμμές οι οποίες φέρνουν ε, τα εμπορεύματα σε αρτηρίες. Εγώ θα επανέλθω στην Κομισιόν, θα ρωτήσω για ποιες από τις οδούς αυτές πρόκειται για το Ευρωβελό απήντησε ο κ. Κουμουτσάκος. Ο κ. Σάβησα επίσης είπε κάτι σχετικά. Εμείς θα επανεξετάσουμε recital και κείμενο. Εμείς έχουμε ρίξει ιδιαίτερα το βάρος μας πρώτα στο νομοθετικό κείμενο. Θα επανέλθουμε και στην σωστή διατύπωση μεταξύ recital, δηλαδή σκέψεων δηλαδή, και κειμένου. Ο κ. Μπενιό μίλησε για τον συγχρονισμό των συνδρομικών δικτύων με τα Cornet και αυτό μας απασχολεί. Αναζητούμε τώρα ένα ξεκάθαρο ορισμό για το τι θα σημαίνει αυτός ο συγχρονισμός. Τελειώνοντας, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο Σίμψον που έθιξε ξανά το θέμα και ευχαριστώ και ζητώ μάλλον ε, την κατανόησή σας ότι δεν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κατάλογος με περιφερειακές επιθυμίες. Γνωρίζω ότι και η πίεση είναι μεγάλη και η επιθυμία είναι έντονη, αλλά ήδη έχουμε περίπου εξαντλήσει τα όρια της ευελιξίας που διαθέταμε. Προσπαθήσαμε να καταστήσουμε δυνατόν κάτι, κάθε που ήταν δυνατόν να γίνει δεκτό αλλά πρέπει να είναι νομοθεσία που να διαθέτει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Αυτό είναι ο προσανατολισμός μας και δεν θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε, κύριε Σίμψον, να γίνει απλά ευχολόγιο ή κατάλογος χριστουγεννιάτικων ονείων. Είμαι στη διάθεσή σα, βέβαια και τις επόμενες δύο εβδομάδες ε, είμαι στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Ερτούκ. Παρατηρήσει κύριε Σέντερ χωρίς μικρόφωνο. Well, Μήπως είναι καλύτερο να τα πείτε μεταξύ σας. Πέστε τα μεταξύ σας. Βεβαίω είναι πάντα σημαντικά όλα όσα ε, έχουμε να πούμε. 18 Δεκεμβρίου και προγραμματισμός είναι για να πάει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου, ενδεικτικός βέβαια. 18 Δεκεμβρίου πρώτα. Ευχαριστώ όλες και όλους. Ευχαριστώ τους κοιόδης, τους συνεισηγητές που μας κατήφθηναν, μας έδειξαν τον δρόμο δηλαδή και το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η είναι το τμήμα τρίτο ε, σχέδιο γνωμοδοτήσεως για το γενικό προϋπολογισμό. Κυρία Ντυρόν. Πριν αρχίσεις, Ιζαμπέλ, όσοι αποχωρούν, να αποχωρήσουν ησύχω, παρακαλώ, και τα πηγαδάκια εκτός αίθουσας. Άρα διαδικαστικό προηγουμένως, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να καθυστερήσω τη συζήτηση περισσότερο, αλλά δεν θα βοηθούσε και με άλλους συναδέρφους, γιατί η απαλλαγή της Επιτροπής και των υπηρεσιών οργανισμών είναι θέματα συνδεδεμένα. Οπότε μήπως να κάνουμε τη συζήτηση ως κοινή αφού προηγουμένως παρουσιάσουν οι συγητές τις γνωμοδοτήσεις τους. Ευχαρίστως. Λέω ο Πρόεδρος, εφόσον συμφωνούν και τα μέλη της Επιτροπής μας, ναι. Συμφωνείτε και εσείς και Μίσνερ, να ακολουθήσετε μετά την κυρία Ντουιρό. Συμφωνείτε? Καλώς τότε. Ωραία. Ιζαμπέλ, αρχίζεις εσύ για τον προπολογισμό και μετά Τζεσίν Μέισνερ θα ακολουθήσει. Ναι, ναι. Ευχαρίστως και πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω το σχέδιο αυτό απαλλαγής προς την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού για το 2011. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για ταχύτητα με την οποία δούλεψαν, έκαναν ό,τι έπρεπε. Απλώς θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία θα έχετε διαβάσει βέβαια το κείμενο και βλέπετε, συζητάμε πάρα πολύ για τη σχέση των υποχρεώσεων και των πληρωμών στον προπολογισμό. Λοιπόν, στο σημείο 5 πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μια χρήση 100% των υποχρεώσεων και 98% των πληρωμών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο κείμενο όμως προτείνουμε από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προπολογισμού για να τηρηθεί αυτή η προσπάθεια της Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικά Κοινοβούλια συνδεόμαστε πάρα πολύ εθνικοί προπολογισμοί δηλαδή με τον ε, Ευρωπαϊκό. Δεύτερον, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία λεπτομέρεια όσον αφορά το επίπεδο πιστώσεων και τη χρήση του το 2011 για την ασφάλεια στις μεταφορές. Ενώ η ασφάλεια είναι κάτι ζωτική σημασία και με εκπλήσει ειλικρινά που δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το γιατί. Και το τρίτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το ποσοστό ε, χρήσης είναι πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τον ε, τουρισμό στην Ευρώπη και είναι καλό αυτό γιατί κάναμε σύσταση εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Τώρα πρέπει να υπάρξει ένα πολιετές ε, πρόγραμμα για τον βιώσιμο τουρισμό. Οπότε με το κείμενο αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει, να προτείνει ένα πολιετές πρόγραμμα για έναν βιώσιμο τουρισμό. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε την απαλλαγή στην Κομισιόν με τις παρατηρήσεις βέβαια που είναι εδώ γραμμένες αλλά και με αυτές που σας ανέφερα προφορικά. Ευχαριστούμε. Κυρία Μάισνε τώρα για τους οργανισμούς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης της κυρίας Γκυρών. Να πω πρώτα τα σχετικά και μετά για τους οργανισμούς. Για την κυρία Ντιουράν συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε. Και θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Αφενό βρίσκω σωστό ότι γίνεται έκκληση στι χώρε μέλη για τα 10T, ώστε να εξασφαλιστούν οι εθνικές χρηματοδοτήσεις. Αυτό έχει κέρια σημασία και αυτό, γι' αυτό παλεύουμε και στην ε, διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη και για τον τουρισμό το ίδιο, να υπάρχουν δηλαδή πολιετή προγράμματα. Τώρα, οργανισμοί. Πρώτα, έμσα όπως είναι και το σχέδιο ΕΜΣΑ Απαλλαγή να δώσουμε, οπωσδήποτε, το λέω ήδη από την αρχή. Κάτι που με εξέπληξε είναι επειδή η ΕΜΣΑ έχει αναλάβει πολλά καθήκοντα, τα οποία είναι και σημαντικά. Περίπου 5% των θέσεων δεν έχουν καλυφθεί. από τις 208 νομίζω έχει μόνο ε, καλυμμένες 190 περίπου. Το ίδιο σημαντικό για το μέλλον, εφόσον αναλάβει περισσότερα καθήκοντα, πρέπει η χρηματοδότηση να είναι εξασφαλισμένη. Και σημαντικό είναι επίσης η Κομισιόν, και γι' αυτό το επαναλαμβάνω εγώ, να κάνει μια πρόταση για την χρηματοδότηση των πολιετών προγραμμάτων του οργανισμού για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρήπανσης. Αυτά για την ΕΜΣΑ. ΕΑΣΑ τώρα, και εδώ είμαι γενικώ υπέρ της χορηγήσεως της απαλλαγής. Εδώ επισημαίνω ιδίω ότι η Άσα σημειώνεται στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων. Η ΑΣΑ δεν έχει κώδικα διοντολογίας για τα θέματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει ας πούμε εργαστεί ε, στην Airbus μετά να αξιολογείται για να εργαστεί στην ΕΑΣΑ. Το ελεγκτικό συνέδριο είχε εξετάσει διάφορους οργανισμούς και τους χειρότερους βαθμούς έβγαλε η ΑΣΑ. Το καλό είναι ότι αντέδρασε γρήγορα και είπε ότι έχουν τώρα κώδικα δεοντολογίας, θα κάνει και σχετική εκπαίδευση. Έχουν δε ήδη τα ηγετικά της τελέχη καταθέσει τις ε, ετήσιες δηλώσεις τους ε, οικονομικών συμφερόντων. Άρα είναι σαφώς βελτιωμένα τα πράγματα και η ΆΣΑ όπως και η ΕΜΣΑ είναι σημαντική όπως η ΕΜΣΑ για την ε, θαλάσσια ε, ασφάλεια η ΆΣΑ για την ε, ενέργεια. Τώρα, ΣΕΣΑ πρώτα όμως ο οργανισμός των σιδηροδρόμων το πιο περίπλοκο πιο περίπλοκος οργανισμός πέρσι είχαμε διστάσει να χορηγήσουμε την απαλλαγή και κυρίω λόγω μεταφορών από παρελθόντα έτη. Ωστόσο, στο μεταξύ έχουν γίνει βελτιώσει, έστω και αν η εικόνα δεν είναι απολύτω ικανοποιητική ακόμα. Είπαμε πως πρέπει να τους, δείξουμε την κίτρινη κάρτα. Πάντως η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του οργανισμού. Βέβαια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων παίζει κέριο ρόλο για την, στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου χωρίς σύνορα. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με ποιον τρόπο εξελίσσεται η διαδικασία. Εφόσον δεν τηρείται η αρχή του ετησίου του προϋπολογισμού. Όμως, όπως είπα, υπάρχει κάποια βελτίωση. Τέλος, η ΣΕΖΑ, σύντομα, προκειμένου, είναι σημαντικός οργανισμός αυτός, για το σύστημα διαχείρισης του ενέργειου χώρου. Πάλι εδώ καλύπτονται μόνο οι 34 από τις 39 οργανικές θέσεις. Και εδώ λοιπόν υπολείπεται ένα 10% περίπου. Μήπως δεν υπάρχει πολλή δουλειά, γι' αυτό δεν ε, προσλαμβάνονται αρκετοί. Είναι σημαντικό ο κοινό ενέργειο χώρο. Αλλά πώ είναι δυνατόν να μην καλύπτονται 10% των οργανικών θέσεων. Κατά τα άλλα είναι εντάξει τα πράγματα και το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε εντάξει τους οργανισμούς και μπορούμε να προτείνουμε χορήγηση τη απαλλαγή. Ευχαριστώ. Άρα, είπατε, ΣΕΣΑ πάτε να βγάλετε την κίτρινη κάρτα, αλλά μάλλον όχι. Και για την αίρα τους έχετε δώσει τον, την κίτρινη κάρτα καλά. Ο κ. Ρικέ από το Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το συγγνώμη Εξ ονόματος του σκιώδους εισηγητή μας, ε, του κυρίου Νταντάν, που αυτή τη στιγμή ως εισηγητής για την κοινή γερική πολιτική ε, είναι πολύ απασχολημένος και έτσι δεν μπόρεσε να είναι εδώ. να αφορά την απαλλαγή για την ε, Κομισιόν, ε, ο σκιώδης εισηγητής θέλει να στηρίξει την απαλλαγή και προκύπτει από την εξέταση του, του Ελληνικού Συνεδρίου ότι ένας βασικός κίνδυνος κανονικότητας είναι ότι η δεν εντοπίζει αρκετά ε, καιρός ορισμένα προβλήματα. Να μιλήσουμε και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη σεβασμού της ε, κανονικότητας. Έχουμε εδώ προσθέσει τις σχετικές κυρώσεις. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να περνάνε τέτοιου είδους ε, παρατυπίες ε, που ε, μάλιστα μια περίοδο που κάθε τελευταίο ευρώ ε, μετράει. Το είπε και η κυρία Ντυρό, θα πρέπει οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται καλύτερα στις μεταφορές. Έχουμε φορείς επιτόπους που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα χρήματα που απελευθερώνονται για την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων. Υποστηρίζω επίση την κυρία Ντουράνο μιλά για την βιοβούληση των κρατών μελών για ικανοποιητικό και εκτέλεση του αν το Συμβούλιο συνεχίσει σε αυτήν την αντιευρωπαϊκή του πορεία, δεν θα μπορέσουμε να προκαλέσουμε τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Χρειάζεται λοιπόν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια να απορροφηθούν από τους δικαιούχους. Ωστόσο, ε, ε, συμφωνούμε για την απαλλαγή της Κομισιόν για την εκτέλεση του προπολογισμού ε, δεύτερη απαλλαγή για τους οργανισμούς. Ο σκιώδης εισηγητής μας θα ήθελε καταρχήν να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την εργασία της στις διάφορες εκθέσεις όσον αφορά την απαλλαγή των διαφόρων οργανισμών, απαλλαγή που δεχόμαστε να δώσουμε για όλους τους οργανισμούς γιατί οι λογαριασμοί θεωρήθηκαν όλοι, κρίθηκαν όλοι αξιόπιστοι. Να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να θυμίσουμε ότι θέλουμε, αν θέλουμε να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες των οργανισμών όπως κάναμε για την ΕΜΣΑ, ε, και μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να οδηγείται η Κομισιόν για τον Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Οργανισμό στη πρόταση για το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Είναι επιτακτική ανάγκη να, γίνει, να υπάρχει ο κατάλληλος προπολογισμό γιατί ένας οργανισμός χωρίς κονδύλια δεν είναι αξιόπιστος ε, και θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανονισμοί που έχουμε φτιάξει. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο διευκολύνεται μέσω αυτών των οργανισμών και να προσθέσω δύο λόγια ότι όπως κάθε χρόνο εμείς κραδένουμε την κίτρινη κάρτα για τον συνδρομικό οργανισμό όμως να θυμίσω ότι ακόμα ανηφόρα ανεβαίνει αυτός ο οργανισμός γιατί υπάρχει μια διαφορά στην εκτέλεση του προπολογισμού την ετήσια έχει φτάσει τώρα στο μάξιμο που της έχει δοθεί είναι σχεδόν δηλαδή στην ρύθμιση πια στην ε, και κατά κάποιο τρόπο δηλαδή φτάνει στην κατάλληλη φάση και να μην την ε, ε, αποδυναμώσουμε γιατί θα τη ζητήσουμε μάλλον περισσότερα μέσα στο πλαίσιο του τέταρτου πακέτου. Ζητώ λοιπόν μια κάποια επίοικια, το βαθμό που η τάση είναι, η πορεία είναι καλή, έχει προχωρήσει και θα τη χρειαστούμε. Δεν βλέπω λόγο να μην δοθεί λοιπόν η απαλλαγή. Τέλο. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο για του περισσότερου οργανισμούς ε, είπε ότι η διαδικασία επιλογής δεν ήταν απόλυτα διαφανή. Στο σημείο αυτό ελήφθη υπόψη από τους οργανισμούς και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου ως προς αυτό. Η σύσταση λοιπόν του κυρίου Νταντάν, του σκιώδη είναι να δοθεί απαλλαγή σε όλους τους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ. κυρία Αγιάλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ. Εκ μέρους της σκιώδους εισηγητριάς μας, της κυρίας Σίδερ. Για λόγους δημοσιονομικούς ακριβώς έχει άλλη, άλλες υποχρεώσει. υποχρεώσεις. Βασικά συμφωνούμε λοιπόν και εμείς με την ε, απαλλαγή όσον αφορά τις μεταφορές Εξάλλου από αυτά που ακούσαμε και από την κυρία Τουράν και από την κυρία Μέσνερ είναι σωστοί λογαριασμοί. Όμως για το Μάρκο Πόλο ίσως θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε την άποψή μας μέσω μιας τροπολογίας για παράδειγμα ότι ελπίζουμε στο μέλλον να λυθούν με την νέα προγραμματική περίοδο τα θέματα αυτά. Και όσον αφορά για το ΣΕΣΑΡ, και στο κείμενο της κυρίας Μέισνερ θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε κάτι που αναφέρεται στο σημείο 4 της γνωμοδότησης της κυρίας Ντουραν που κάνει μια σύνδεση με την αλλαγή στη μεθοδολογία και να αναφερθούμε στα προβλήματα του οργανισμού της ΕΑΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όλοι οι οργανισμοί, φαίνεται και στην έκθεση Κεμπραντή από την Κοκομπή, εγώ είμαι ότι πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας ε, δεοντολογίας. Στο κείμενο για την Ιάσα λέει ότι είναι ένα θέμα για την ασφάλεια της αεροπλοίας. Άρα επήγει πιο πολύ, αλλά και για τους άλλους οργανισμούς κάποια στιγμή θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας κώδικας δεοντολογίας όταν δημιουργούνται ε, προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα. Πάντως, χρησιμοποιήθηκαν ε, καλά τα χρήματα για τον τουρισμό και άρα να ενισχυθεί αυτό που λέμε και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Έτσι, όπως έχουν οι νέες προτάσεις, όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να λυθεί το θέμα της πλατφόρμας. Όσον αφορά για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, χαιρετίζουμε τις δυνατότητες που έχουν και σε σχέση με τα μελλοντικά καθήκοντα, στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, ελπίζω να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε. κύριος σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω να κλείσει αυτή η ιστορία και να μην καθυστερήσουμε, αλλά δυστυχώς έχω να πω αρκετά πράγματα. Εν γέννη ήθελα να πω, γιατί φαίνεται ότι κανείς δεν το, να μην το αναφέρει, ίσως και να μην το έχει διαβάσει, ότι στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό, στην έκθεση μάλλον του Ευρωελεκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση του περσινού προϋπολογισμού και πάλι για 18η χρονιά δεν έχει δώσει το πιστοποιητικό ε, ξεπιστίας και αν μη τι άλλο αυτό προκαλεί ερωτήματα ιδιαίτερα για τα θέματα με τα οποία εμείς ασχολούμαστε εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει λέμε πως έχουμε ποσοτικά ότι οι λογαριασμοί έχουν υπογραφεί, αλλά τι γίνεται με τους, τις ποιοτικού όρους. Και αν δούμε την έκθεση που έχουμε μπροστά μας τώρα, όπου οι μεταφορές ε, έχει, συνοψιστεί με την ενέργεια και την περιφερειακή πολιτική, με εντυπωσιάζουν οι συναλλαγές εδώ. 59% των συναλλαγών έχουν σφάλμα. Αυτό είναι εξοργιστικό. Πώς χρόνο με το χρόνο μπορούμε να είμαστε εδώ και να επικρίνουμε και να επικρίνουμε και στο τέλος ό,τι και αν λέμε ναι τελικά άντε ας δώσουμε την απαλλαγή. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Να μπω τώρα στο θέμα των οργανισμών. Συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Μάιζνερ για την ΙΑΣΕ και για την ΙΑΡΕΗ ε, Όχι πάλι, ούτε καν κίτρινη κάρτα. του έχουμε δώσει κίτρινε κάρτε εδώ και καιρό. Τώρα πια κόκκινη κάρτα πρέπει να τους ε, δείξουμε. Θυμάμαι, δεν έχω βέβαια τα στοιχεία τώρα μαζί μου όσον αφορά την Ιάση, αλλά θυμάμαι πως το συζητούσαμε εδώ στην Επιτροπή για το τεράστιο διοικητικό κόστος του οργανισμού αυτού σε σχέση με την αναλογία και τον γενικό του προπολογισμό. Τι έχει γίνει για να κατεβεί το κόστος στο διοικητικό. Γιατί οι εταιρείε ξέρουν να το πληρώνουν αυτό μέσω των ε, ε, τελών που χρεώνει η ΆΣΕ. Και θυμάμαι ότι έχουμε επανέλθει για τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά ένα διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θυμάμαι να πήραμε ικανοποιητική απάντηση και για την ΕΡΑ πάλι ναι, σωστά Ξεκολουθούν να υπάρχουν ζητήματα εκκρεμή. Αν εν γέννη βλέπουμε αυτούς τους οργανισμούς, πρόκειται για περίπου 10.000 κόσμο που απασχολείται σε αυτούς τους οργανισμούς, αλλά ποτέ δεν βλέπουμε κανένα σημάδι μείωσης, ε, αντίστοιχης μείωσης προσωπικού στην Κομισιόν, που υποτίθεται ότι ανέθεσε αυτή τη δουλειά που έκανε στον εκάστοτε οργανισμό. Στην ουσία αντιστρέφεται η τάση που εξακολουθεί εδώ και κάποια χρόνια, ότι δηλαδή προσπαθούμε όλα αυτά να τα κάνουμε καλά, αλλά τελικά μάλλον λάθος πάντα πράγματα. Δεν διορθώνεται τίποτα. Εγώ λοιπόν, Πρόεδρε, φοβούμαι πως, κλείνοντας, εγώ δεν μπορώ να βρω καμιά λογική να συνεχίσουμε τις κριτικές και τις επικρίσεις και μετά από όλες αυτές να ξαναδίνουμε την απαλλαγή. Εγώ δεν πρόκειται να τις υπερψηφίσω αυτές τις απαλλαγές. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τους οργανισμούς εν γέννη, τα προβλήματα είναι διαφορετικά από τον ένα οργανισμό στον άλλον. Έχουμε το πρόβλημα των περιστρεφόμενων ε, θυρών. Χρειαζόμαστε δηλαδή εμπειρογνώμονε που να είναι εμπειρογνώμονε, αλλά να είναι και ανεξάρτητοι και σε πολλέ από τι δηλώσει που ακούμε, τι επικρίσει, τι παρατηρήσει κτλ. Ε, βέβαια όλα αυτά τα λέω με ιδιαίτερη προσοχή αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο που εργάζεται στη σιδηροδρομική ε, οργανισμό, στον οργανισμό σιδηροδρόμων ή στην ΕΑΖΑ μπορεί πραγματικά να αρνηθεί την αρχική του εκπαίδευση και το αρχικό του επάγγελμα και αυτό το πρόβλημα το διαπιστώνουμε σε διάφορους οργανισμούς είναι όμως πολύ σοβαρό γιατί πρέπει να λάβουμε ευρωπαϊκές προσεγγίσεις, να ακολουθήσουμε ευρωπαϊκές προσεγγίσεις που να μην αφορούν μόνο κάποιους τομείς του κλάδου. Το πρόβλημα αυτό είναι μεγάλο και έχει μεγάλο κόστος αξιοπιστίας. Γι' αυτό και πρέπει οι οργανισμοί να το λάβουν πολύ πολύ εντονότερα υπόψη τους. Σαρβάμα. Σαρβάμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης του Λαϊκού Κόμματος για τις απαλλαγές αυτές θα ήταν χρήσιμο για μένα να ακούσω λίγο περισσότερο από την κυρία Μάισνερ. Αυτά που είπε ο κύριος Μπράντμπουν με απασχολούν και εμένα. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι εν τέλει τι σας έπεισε εν τέλει, γιατί και εσείς είπατε στις παρατηρήσεις σας ότι ο ERA ήταν πέρσι ο πιο προβληματικός οργανισμός. Και σχεδόν είχατε καταλήξει να τους δείξετε την κόκκινη κάρτα και φέτος όχι. Δεν προσπαθώ εδώ να ε, πω κάτι ιδιαίτερο, αλλά θα ήθελα να μάθω ποια ήταν τα γεγονότα που σας έπεισαν φέτος ότι ο οργανισμός για τους ιδιοδρόμους δεν είναι πλέον τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο ήταν πέρσι. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, να πω το εξή, λέει ο Πρόεδρος. είναι η επάνδρωση. Και ο τρόπος διορισμού των στελεχών αυτών. Κάπως μου φαίνεται σαν ένα κλειστό κύκλωμα για το ποιοι παίρνουν τις δουλειές αυτές. Κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και την εμπειρία είτε διότι έχει εργαστεί σε σιδηρόδρομο ή σε αεροπορική εταιρεία. Είναι καλύτερο παρά να πάρουν, για το που έτσι, χονδροειδός κάποιον από το κτίριο Μπρελεμό και να τον βάλουν στον οργανισμό. Αυτό με απασχολεί. Λοιπόν, ο κ. Τόσμαν της Κομισιόν. Έχετε ένα οργανισμό με κίτρινη κάρτα έναν οργανισμό που σκεφτόμαστε να του δώσουμε και κάρτα και μερικές ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο που προσλαμβάνονται ή δεν προσλαμβάνονται ε, μέλη του προσωπικού. Εσείς έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ στους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές ε, για την γενικά ε, θετική άποψη που έχετε, καθώς επίσης ευχαριστώ και για τις κριτικές σας διότι βέβαια τα θέματα που θέτεται δεν είναι και άγνωστα σε μας. Ας πάω όπως πήγε ήδη η συζήτηση, μια σύντομη παρατήρηση για το γενικό προϋπολογισμό και μετά να εξετάσουμε από κοντύτερα τους οργανισμούς και να σας δώσω ορισμένες εξηγήσεις ή εν πάση περιπτώσει κάποια εισφορά στη συζήτηση. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την υπόψη την γνωμοδότηση κ. Ντυράν. Προετών το 2009 είχαμε αρχίσει με πολύ υψηλέ ε, απαιτήσει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ή των μεταφορών μάλλον, το 2009. Το 10 και 11 πήγαμε, ε, πήγαμε στα 86 και 95 και σας εξηγήσαμε τι κάναμε με τα σχετικά κονδύλια και συνεχίζουμε. Παραμένουν αυτά δηλαδή, τα έχουμε αυτά από υπόψη μας. Τώρα, για τους οργανισμούς, για την ΕΜΣΑ, εξηγήσατε το δίλημα και εν μέρη την απάντηση σχετικά με το τι γίνεται με τις κενές θέσεις. Τα όργανα μας γενικά, Κομισιόν, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο 2-3% κοινέ θέσει είναι λίγο πολύ κανονικέ. Διότι κάποιοι φεύγουν, πρέπει να αντικατασταθούν, αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Για την ΕΜΣΑ λοιπόν έχουμε αυτό το 5%. Και μετά για την ΣΕΣΑ στο υψηλότερο ποσοστό που σημειώσατε. Το 2% παραπάνω από τον μέσον όρο έχει σχέση με το ότι πρόκειται για πολύ εξειδικευμένες θέσεις και είναι δύσκολο καμιά φορά να προσληφθούν πρόσωπα σε συμπαθητικούς αλλά όχι πολύ κεντρικούς ευρωπαϊκούς τόπους. Αυτό το 5% βέβαια θα πρέπει να μειωθεί, όντως. Αλλά πρόκειται για πολύ εξειδικευμένες θέσεις. Το άλλο πράγμα που βλέπει κανείς στον, στη ζωή ενός οργανισμού είναι ότι προσλαμβάνονται σε δεδομένες χρονικές στιγμές κάποιες ομάδες ανθρώπων με συμβάσεις. Αυτοί, ε, οι συμβάσεις αυτές λήγουν σε μια πενταετία συνήθως και γι' αυτό υπάρχει μετά ένα κενό, μια διακύμανση. Κάτι το οποίο δείχνει σαν να είναι ανισχυτικό, αλλά στην πραγματικότητα θα καλυφθεί το κενό αυτό. Βέβαια, ειδικά για την ΣΕΣΑ, θα επανέλθω, θα έλθω σε επαφή με την αρμόδια μονάδα σε εμά, γιατί βέβαια το 10% ε, έχετε δίκιο είναι πολύ υψηλό για να λειτουργήσει σωστά ο οργανισμός. Για τον ΕΜΣΑ, το γεγονός, το θετικό είναι ότι η πρόταση για την πολιτική χρηματοδότηση είναι έτοιμη, θα προχωρήσει στην διαδικασία εγκρίσεως και θα σα υποβληθεί. Για την ΙΑΣΑ λέτε σωστά και το σημειώνουμε ότι μετά από τα προβλήματα τα οποία αναφύγηκαν αναλύθηκε δράση και από τον οργανισμό αλλά και από την Κομισιόν. Για όλους τους οργανισμούς άλλωστε, γιατί εγώ είμαι αρμόδιος και για την ενέργεια, η διαθεσμική προσέγγιση που εγκρίνατε εσείς μαζί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν βοηθεί πολύ για να υπενθυμίσουμε στους οργανισμούς τους βασικούς κανόνες που διέπουν τις εργασίες τους και εν πάση περιπτώσει ο δικό μας τομέα το περνάμε το μήνυμα σαφέστατα και με αιμονή στους διάφορους οργανισμούς. Για τον ERA συμφωνώ με την άποψη ότι κάποια στιγμή το 100% των δαπανών για το συγκεκριμένο έτος πρέπει να πληρώνει το συγκεκριμένο έτος. Ο ΕΡΑ, ωστόσο, βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Πλησιάζουν τώρα, θα έλεγα, ένα ικανοποιητικό ή και εξαιρετικό ρυθμό εκτελέσεων. Και νομίζω έχουν κατανοήσει και στον οργανισμό την ανάγκη αυτή και θα έχουμε καλύτερα νούμερα του χρόνου. Γενικά βεβαίως η συζήτηση αυτή είναι εκτενέστατη. και είπατε και εσείς πρόεδρε τι γίνεται, πώς είναι δυνατόν να αυξάνει το προσωπικό των οργανισμών και αν μειώνεται το προσωπικό των Κομισιόν. Στο σχέδιο προπολογισμού του 2013 η Κομισιόν σημειώνει ότι η συνολική μείωση του προσωπικού κατά 1% εφαρμόζεται και στους οργανισμούς. Και έχει προταθεί αυτό, αυτούσιο. Και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις εσωτερικά στην Κομισιόν, εάν αυτό είναι πάντοτε δικαιολογημένο. Στο τέλος όμως θα δείτε ότι όλοι οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το σενάριο το οποίο καλώς γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντυρά. Θέλετε εσείς πρώτα να πάρετε το λόγο και μετά η κυρία Μέσνερ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις που έκαναν οι Σκιώδης και για τόσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα για τις δαπάνες στον τομέα της ασφάλειας που αυξήθηκαν αλλά, για το μέλλον δηλαδή, αλλά εδώ μιλάμε για την απαλλαγή για το 2011. Οπότε την απαλλαγή αυτή συνολικά πιστεύω ότι μπορούμε να τη δώσουμε στην ε, Κομισιόν. Αλλά οι παρατηρήσεις των συναδέρφων στέκουν σίγουρα. Το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων έχει μεγάλη σημασία για τους οργανισμούς και είναι καλό να έχουμε πραγματογνωμοσύνη εκτός ε, των οργανισμών. Αλλά δεν υπάρχει μόνο τον Περλεμόν γι' αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα στην απαλλαγή που δίνουμε. Για μένα είναι ζωτική σημασία για το μέλλον. Το έχουμε δει και σε άλλους οργανισμούς. Εκείνη για την ασφάλεια των τροφίμων, για παράδειγμα. Θα τα θυμόσαστε τώρα αυτά που έχουμε πει. Καλύτερα η πρόληψη λοιπόν παρά η θεραπεία. Ευχαριστούμε. Συζήν. Επί των όσων ελέγχθησαν, λίγο πολύ νομίζω ότι με στηρίζουν στα όσα είπα. Βέβαια, η ανεξαρτησία είναι απόλυτα σημαντική. Κανένα δεν την πετύχει ποτέ 100%, αλλά αυτό πρέπει να είναι ο στόχο μα. Και έτσι είναι σημαντικό να διαθέτουμε του οργανισμού αυτού και να λειτουργούν. Τώρα, για ό,τι αφορά, ό,τι αφορά τον ΣΕΖΑ. Κρίμα που η Κομισιόν δεν μπορεί στην πραγματικότητα να μα πει γιατί υπάρχει αυτό το κενό των 10%. Εάν πραγματικά δεν είναι απαραίτητε αυτέ οι θέσει, τότε ίσω πράγματι να πρέπει να δούμε μήπως μπορούν να εξοικονομηθούν. Εάν μας προβάλλουν την αιτιολογία ότι χρειάζονται λόγω του European Sky, τότε ναι. Αλλά είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι δεν έχουν επανδρώσει τις θέσεις εφόσον δεν τις χρειάζονται. Για τον σιδηροδρομικό οργανισμό. Δίστασα διότι ήμουν πέρσι και σκιώδης συγγήτρια και είπα ότι όταν βλέπουμε να μη λαμβάνουν υπόψη το ετήσιο του προπολογισμού και να κάνουν μεταφορές κονδυλίων, αυτό πρέπει να σημειωθεί. Τώρα βέβαια κάποια βελτίωση υπήρξε. Το ότι προτείνω απαλλαγή έχει σχέση με το γεγονός, όπως είπε και ο κύριος Ρίκη, Ρικέ μάλλον, για το τέταρτο πακέτο των σιδηροδρόμων, η Κομισιόν θα αναλάβει Α, ο οργανισμό εννοώ που είναι σημαντικό για την Κομισιόν, ωστόσο, αν λαμβάνει περισσότερα καθήκοντα. Μα τότε λέω εγώ ότι πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι λειτουργεί λογικά σωστά. Ανεξαρτήτως του τι θα πράξω εγώ του χρόνου, θα εξετάσω πάντω πολύ προσεκτικά τον οργανισμό αυτό και την λειτουργία του. Πάντως, εν τέλει, εγώ προτείνω τη χορήγηση της απαλλαγής. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. Ιδιαίτερα για τις θέσεις που καλύπτονται. Εγώ πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία πρόσληψης. Γιατί η Επιτροπή έχει τα δικά της κριτήρια τα οποία εξάγονται στους οργανισμούς για να καταλήξουν στο ποιος είναι ο καλύτερος να πάρει την κάθε θέση. Το έχουμε ξαναδεί το πρόβλημα αυτό. Αν δεν μιλάς 37 γλώσσες, για παράδειγμα, μπορεί να είσαι ο καλύτερος μηχανικός γενικής για παράδειγμα, αλλά δεν ε, κάνεις. Θέλεις δηλαδή και τους εμπειρογνώμονε και τις γλώσσε. Εγώ λέω ότι θες του εμπειρογνώμονε για τη συγκεκριμένη δουλειά και όχι αυτούς που μιλάνε τι 37 γλώσσες. Αυτό είναι το θέμα. Θέλουμε ειδικού επιστήμονες, ναι, ανεξάρτητους. Ωραία. Καλώς. Τον Ιανουάριο θα ψηφίσουμε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 12η Δεκεμβρίου. Στις 12 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Καλώς. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη τώρα. Εντάξει, αφού φτάνει θα το προχωρήσω γιατί αν κάνουμε διάλειμμα δεν θα ξανάρθουν, για τις ε, κατεξοδότηση πράξεις. Is that the commission? Philip's having the 10 minute break anyway. Ο Φίλιπ το κάνει το δεκάλεπτο διαλυματάκι του, ούτως ή άλλως. If there's a, I mean, it was scheduled at 5, I don't know why they are not Okay, well, I'll just, I will have to wait for the commission to... Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 5 τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, οπότε αναγκαστικά μάλλον θα μου δώσω την έκθεση, αλλά 15 λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ. Okay, colleagues, the commissioner's arrived. The next item on the agenda. Εντάξει, συνάδελφοι, έφτασε εκπρόσωπο του Ισ Επόμενο θέμα είναι η πρώτη κατεξοδότηση πράξη για την οδηγία ITS Equal από την Γενική Διεύθυνση MOVE. Πρόκειται για την πρώτη κατεξουδότηση πράξης ε, που εμπίπτει στην ε, εντολή της, εποστο... της... Ε, της Επιτροπής μας, εναρμονισμένη δηλαδή διάταξη για το e call για τα FEE συστήματα μεταφορών. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η συντονισμένη ανάπτυξη και χρήση εφιών συστημάτων μεταφορών στους, στις οδικές μεταφορές ολόκληρη την Ευρώπη. Άρθρο 7 αυτές τις οδηγίες ε, επιβάλλει στην Κομισιόν να υιοθετήσει την κατοξιδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 219 της ΤΕΦΙΓΙΟ όσον αφορά τις συγκεκριμένες ε, δράσεις προτεραιότητας. Η κατεξιδότηση πράξη αποτελεί επίσης ε, το σημείο ενημέρωσης ε, της δημόσιας ασφάλισης, τη, δομή, τη σχετική δομή της Κομισιόν, πράγμα που έχει οθετήσει σε πρόσφατη έκθεσή του το Κοινοβούλιο, ε, έκθεση που υπέβαλε η κυρία Σαβαλόβα της ΣΥΜΚΟ και ο κύριος Κότ θα ευχαριστώ, την Ευρωπαϊκή Κομισιόν που ήρθε να παρουσιάσει την κατεξοδότηση πράξη και τη συνεργα... πνεύμα συνεργασία που έδειξαν κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία τη πράξη αυτή. Είχαμε εντατική ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις επαφές με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες για την προετοιμασία των όλων των στοιχείων εκεί όπου έχει προσκληθεί και η Επιτροπή Μεταφορών. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και μετά θα ακούσουμε με το, θα δούμε μάλλον με τα μέλη ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν έχω το όνομά σας, συγγνώμη. Ε, πείτε μας το όνομά σας, παρακαλώ, συστηθείτε. Ολιβιέ Ονιντή, από την DG Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ πρώιμη ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε αυτήν την πρώτη κατεξοδότηση πράξη που προτείνεται υπό την οδηγία για τα ΕΦΗ συστήματα μεταφορών. Η πρώτη αλλά δεν είναι αυτή η οποία δεν, δεν σας είναι άγνωστη γιατί πρόκειται για ένα θέμα και αναφερθήκατε σε αυτό, είναι ένα θέμα επί του οποίου το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγγύψει, έχει ασχοληθεί και έχει δώσει τη στήριξή του. Θα έλεγα ότι μετά από μια χαμένη δεκαετία στην ε, προσπάθεια όθησης του e-call σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση Εν τέλει, ελπίζω τουλάχιστον είμαστε σε μια φάση όπου θα μπορέσουμε γρήγορα να εφαρμόσουμε το e-call. Η συζήτηση αλλά και η πρόταση θα σας φανεί πολύ γνώριμη, διότι <clears throat> ακολουθούμε κατά γράμμα την έκθεση που έχετε εσείς υιοθετήσει τον Ιούλιο. όπως την παρουσίασαν ο κύριος Κόχ με τον οποίο είχαμε την συζήτηση και την κυρία Σαβαρλόβα αυτή η έκθεση είναι η πρώτη από μια τριλογία που θα υποβληθούν, υποβληθεί στην Ευρω... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η έκθεση η οποία φροντίζει το θέμα το υγείας και της ασφάλειας και μάλιστα τις συγκεκριμένες διατάξεις που γνωστοποιούν στις αρχές των κρατών μελών τι είδους προδιαγραφές θα πρέπει να σωματώσουν στα διάφορα συστήματα που υπάρχουν για να μπορέσουν να χειριστούν τα e-calls στην επικράτειά τους. Εδώ εμείς Μιλάμε μόνο για τις απαραίτητες προδιαγραφές, τοποθεσία, κατεύθυνση του οχήματος, ε, τα βασικά στοιχεία του οχήματος και φυσικά την τον οδηγό και τις υπηρεσίες ασφαλείας έτσι ώστε να μπορούν να συνομιλήσουν και να γνωρίζουμε περισσότερα για το ατύχημα ή το περιστατικό. Από τη στιγμή που θα έχουμε τώρα υιοθετήσει τις προδιαγραφές, γρήγορα μέσα στον επόμενο χρόνο θα μπορέσουμε μέσα με μια νομοθετική πρόταση που μάλλον θα είναι οδηγία, να προτείνουμε το τμήμα το εφαρμοστικό. Και με αυτή την οδηγία που τότε θα είναι αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, σε συναπόφαση, θα έχουμε και τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε τις διάφορες διαδικασίες για να μπορέσουμε γρήγορα να εφαρμόσουμε και τις υπηρεσίες. Αυτό ακριβώς είναι που καλύπτεται στην έκθεσή σας που υιοθετήσατε τον Ιούλιο. Να προσθέσω πως βέβαια οι δυο άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργά συνεχίζουν τις εργασίες τους για την Νικόλα. Έχω δίπλα μου τον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση Connect που στενά εξετάζει τα όσα κάνουν οι φορείς το κινητής τηλεφωνίας επί τη βάση των συστάσεων που τους δόθηκαν για να προβλέψουν προδιαγραφές για να μπορέσουν να χειριστούν τις υπηρεσίες e-call και συμπεριλαμβάνει επαφές από την, με την Γενική Διεύθυνση Enterprise. Πιστεύω θα χαρείτε να ακούσετε ότι ολοκληρώνει η DG Enterprise την τροποποιητική νομοθεσία για την έγκριση τύπου που είναι το πιο ορατό τμήμα του Equal γιατί είναι εκείνο το, η νομοθεσία που θα επιτρέψει την λειτουργικότητα και την εσωμάτωση αυτής σε όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ένωση. Με όλα αυτά ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση στις αρχές του επόμενου να έχουμε όλα αυτά τα διαφορετικά τμήματα της νομοθεσίας ε, για το e και θα ξεκινήσουμε πια σε μια επικοδομητική συζήτηση με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο έτσι ώστε πριν το τέλος αυτής της θητείας να έχουν όλα αυτά τεθεί πια σε εφαρμογή. Γιατί είναι ζωτική σημασία σε αυτή η υπηρεσία. Ευχαριστώ. Okay, Mrs. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που δώσατε. Δεν πρόλαβα δυστυχώς να μελετήσω όλο το έγγραφο, όσο γρήγορα και να διαβάζω δεν μπορώ τόσο γρήγορα. Πάντως, για μένα μένουν ανοιχτά ορισμένα ερωτήματα. Πώς μπορεί να αποφευθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα τεχνικό μονοπόλιο. Όταν πρόκειται δηλαδή εδώ για τεχνικές προδιαγραφές θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα ως ένα από τα κέρια σημεία, ώστε να μην υπάρχει ένας όμιλος, ας πούμε, ο οποίος να υποφελείται και οι υπόλοιποι να μένουν εκτός. Δεύτερο, τώρα, από πλευράς υποδομής των χωρών που απαιτείται. Έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν υπάρχουν δυστυχώς πολύ θετικές εμπειρίες. Εάν συγκεντρωθούν όλες ε, οι κλήσεις βοηθείας. Ενδέχεται τελικά να σπεύσουν επί τόπου πέντε διαφορετικές υπηρεσίες όταν υπάρξει ένα τύχημα, διότι είναι ε, λάθος συντονισμός. Ή σε άλλες περιπτώσεις να μην γίνεται τίποτα, διότι δεν λειτουργήσε καλά το σύστημα. Για μένα λοιπόν υπάρχουν ακόμα πολλά ανοιχτά τεχνικά θέματα διαπιστώνετε κι εσείς ότι η μελέτη αντικτύπου είναι δύσκολο να γίνει. Διότι, υποψιάζομαι εγώ, ότι εφόσον γίνει σοβαρά, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που ενδιαφέρουν κυρίως από την πλευρά των υποδομών των χωρών μελών και εκεί οι προδιαγραφές είναι τελώς ασαφείς. Άκουσα ότι σε πιλωτικά προγράμματα και λέω άκουσα, γι' αυτό σας παρακαλώ είτε να το επιβεβαιώσετε είτε να το διαψεύσετε, ότι δεν έχει λυθεί επαρκώς το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, προσωπικών δεδομένων και ότι γίνονται τελικά πολλά, πολύ λάθος συναγερμοί, δηλαδή συμβαίνουν πολλές κλήσεις που είναι λάθος. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα δύσπιστη. Δεν είμαι βεβαία ότι έχει όντως νόημα να προχωρήσετε με τέτοια ταχύτητα. Ένα πράγμα που πρέπει να ρεθεί ακόμη είναι ότι αυτή η συγκέντρωση των υπηρεσιών, για παράδειγμα των υπηρεσιών διασώσεως, σε ορισμένες χώρες μέλη, σε ορισμένες χώρες οι υπηρεσίες διασώσεως είναι εντελώς αποκεντρωμένες και βασίζονται σε εθελοντικές πρόσφορες υπηρεσιών. Αυτά τα χάνουμε με τον τρόπο αυτό. Και αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον τομέα αυτό. Και γι' αυτό η ερώτησή μου είναι, στο impact assessment που έχετε κάνει, έχουν ληφθεί υπόψη αυτά. Έχουμε κάνει εντατικές συζητήσεις για τα συστήματα διασώσεως. Και γι' αυτό σκέφτομαι και νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά, διότι μιλούμε για υποδομές εκατομμυρίων και από πλευράς χωρών όπου τα οικονομικά τους δεν είναι καλά. Βέβαια υπάρχουν και οι εθελοντές είναι σημαντικό όμως σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν ξεκάθαρες προδιαγραφές για την υπηρεσία 112. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάπως πρόωρο λοιπόν στη βάση των υφιστάμενων δεδομένων. Είναι πρόωρο, λέγω, να προχωρήσουμε με νομοθετική ρύθμιση. Με επιβολή δηλαδή νομοθετική ρύθμιση. Κύριε Σεναλόβα, εισηγήτρια της Ήτρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι για την Ήτρε, για την ΗΜΚΟ. Ήμουν συγκήτρια, Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την πρώτη νομοθετική της πρόταση. Πιστεύω ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ομάδα τεχνικών που έχει δουλέψει από τον Οκτώβριο του 2011 πάνω σε αυτό. Οπότε με εκπροσώπους των κρατών μελών συζητιούνται αυτά τα τεχνικά θέματα πολύ έντονα. Έπειτα έχουμε τις προτάσεις επί τάπητος, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με την έκθεση που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καλοκαίρι. Εκεί ζητάμε για το νούμερο αυτό 112 που να εγκριθεί και να μπορούν τα οχήματα να το χρησιμοποιούν και αυτό μέχρι το 2015. Αν θέλουμε όμως να το πετύχουμε αυτό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε την δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με την έκθεση λοιπόν και με αυτά που είπε η κυρία Λίχτεμπεργκ, για το κόστος του μέτρου αυτού στα διάφορα κράτη-μέλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρξει αναρμόνιση βάσει των ε, εθνικών προϋποθέσεων. Και αυτό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας το κόστος και το όφελος το κόστος για τον εξυγχρονισμό των ε, κέντρων που απαντούν πηγαίνει από χίλια μέχρι χιλιάδες και χιλιάδες ευρώ. Αν όμως κοιτάξει κανείς το ωφέλη που θα αποκομίσουμε από το σύστημα αυτό, τα ποσά αυτά ακούγονται πολύ λογικά. Επίσης, το νομοθετικό αυτό βήμα, από ό,τι ακούω, είναι το πρώτο και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Θέλω να υπενθυμίσω επίσης στους συναδέρφους ότι το βήμα αυτό αποτελεί την ενσωμάτωσή του συστήματος μέσα στα οχήματα. Και εξάλλου γι' αυτό και η αυτοκινητοβιομηχανία και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Και τίθεται και θέμα διασυνοριακής διαλειτουργικότητας κτλ. Ήμουνα στην πρώτη διάσκεψη η οποία συζήτησε τα αποτελέσματα στο Ζάγκρε πριν από τρει εβδομάδε. Όλες οι χώρες πρέπει να ξέρετε ότι δουλεύουν εντατικά πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε την προθεσμία του 2015. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε περισσότερο όμως, θέλω να σας πω το εξής. Πώς λειτουργεί αυτή η κατεξουσιοδότηση πράξη πήγε στις 26 Νοεμβρίου, ήρθε μάλλον στο Κοινοβούλιο. Το κείμενο με το σημείωμα που ετοίμασε η Γραμματεία εστάλει στα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Η περίοδος που έχει τώρα στη διάθεσή του για ένσταση το Κοινοβούλιο είναι δύο μήνες που μπορεί να παραταθεί δύο μήνες εφόσον πάρει την πρωτοβουλία το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο η προθεσμία άρχισε να τρέχει από τις 26 Νοεμβρίου. Τώρα, αν ε, κάποιο μέλος Επιτροπής Μεταφορών θέλει η Επιτροπή μας ε, να καταθέσει ψήφισμα στην Ολομέλεια αντιτιθέμενη στην κατάθεση της πράξης, τότε πρέπει να ενημερωθεί η Γραμματεία πριν την 21η Δεκεμβρίου. Γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί μπαίνουμε σε μια συζήτηση πάλι για τα ITS, για τα εφή συστήματα μεταφορών, σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έχει δύο μήνες στη διάθεσή του για ένσταση. Η περίοδος αρχίζει από τις 26 Νοεμβρίου. Συνεπώς, εφόσον θέλετε να κατατεθεί ψήφισμα στην Ολομέλεια, για να αντιταθούμε στην υιοθέτηση της πράξης, τότε πρέπει αυτό να το ξέρουμε πριν από τις 21 Δεκεμβρίου. Η κυρία Μάιστερ τώρα. Ευχαριστώ που το επαναλάβατε. Εμένα μου φαίνεται σαν να ζητούμε ένα δίμηνο παραπάνω. Δεν ξέρω η διαδικασία τι επιτρέπει, γιατί βέβαια μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν είχαμε δύο μήνες Καλύτερα θα ήταν βέβαια αν και είναι στη μέση και οι διακοπές του τέλου του έτους. Τέλος πάντων, αυτό οφείλεται εν μέρει και στο ότι δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο. Ασφαλώς όλοι είμαστε υπέρ των εφιών συστημάτων μεταφορών και απέναντι στο e-call είμαστε επίσης θετικοί. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό ε, σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Για μένα δεν είναι τόσο το θέμα των μονοπωλίων, διότι όταν κάτι το θέλει αγορά, βρίσκονται πολλοί που ενδιαφέρονται. Το ίδιο έχει γίνει και με τα body scanner, μάλιστα αντίθετα με τη βούλησή μας. Και είχαμε πει ότι αφού είναι για τα body scanner θα, τα, θα περιλάβουμε και τα μηχανήματα ακτινογραφιών. Τώρα βέβαια, σε κάθε τεχνολογική καινοτομία αυτό που πρέπει να διασφαλίζεται είναι ότι είναι απλή χρήση της τεχνολογίας και ότι είναι δεδομένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι θέμα βέβαια και των εθνικών μονάδων, αν δηλαδή λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανάγκες τους εφόσον υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Ισχύει και για τη Γερμανία ότι πολλά τμήματα των υπηρεσιών διασώσεως είναι βασισμένα σε εθελοντική βάση Εάν χαθεί αυτό, αυτό θα, είναι, θα έχει το, το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμούμε. Θα είναι ε, κρίμα να χαθούν όλες αυτές οι δυνατότητες που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Τώρα, σήμερα έχουμε 3 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 21 μας μένουν περίπου δύο εβδομάδες. Είναι δύσκολο πώς να αντιδράσουμε σε τόσο λίγο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Για τους δύο έξτρα μήνες πρέπει να μας Γνωρίστε το δυνατόν συντομότερο αν τους θέλετε και να πάει στους συντονιστές να δούμε εάν συμφωνούν να ζητήσουμε τους έξτρα δύο μήνες και να το βάλουμε. Το λέω αυτό για να γνωρίζετε πώς είναι η διαδικασία. Ο κ. Αλχαντράουι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας είναι η συνέχεια που δίνεται σε αυτό που εμείς ως Κοινοβούλιο ζητήσαμε. Εμείς ζητήσαμε νομοθεσία, είχαμε και έκθεση πριν από λίγο καιρό και με αυτήν ζητήσαμε να προχωρήσουμε με τις υποθέσεις αυτές και το ITS. Αυτό είναι το πρώτο. Θέλω να το υπογραμμίσω για να ξέρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα το κείμενο φυσικά πρέπει να το δούμε, να ξέρουμε αν χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Πάντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις κατεξοδότηση πράξεις και την ε, οδηγία που θα ακολουθήσει, που ανακοινώνεται για του χρόνου. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά υπάρχουν έτσι δεν είναι. Δεν θα τροποποιηθούν με την νέα νομοθεσία. Οπότε ρωτάω, ποιος είναι ο στόχος της νομοθεσίας. Είναι θέμα χρονικής στιγμής ή κάτι άλλο. Ίσως η Επιτροπή μπορεί να μου εξηγήσει περισσότερο. Τέλος, υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν και για τη συμπεριφορά διαφόρων χωρών μελών, πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των κρατών μελών επίσης, απέναντι στην πρότασή σας δηλαδή. Ευχαριστώ. The Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα υποβαλώ κανένας είδου ένσταση. Χαίρομαι που επιτέλους προχωρούμε. Έχουμε χάσει μια δεκαετία περίπου. Τώρα, δεν υπάρχει καν λόγος να συζητούμε τον σκοπό. Είναι περιττό. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πραγματικό patchwork. Διαφορετικά συστήματα στις διάφορες χώρες που νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι θετική εξέλιξη κάθε χώρα δηλαδή να προσφέρει την ιδιωτική της λύση. Όπως είπε ο κύριος Σαΐντ, εμείς το έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό. Βέβαια έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη η προστασία δεδομένων, οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαλειτουργικότητα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Πάση θυσία, διότι έχει ήδη απολεστεί πάρα πολύ πολύτιμος χρόνος, η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, γνωρίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά 21 Δεκεμβρίου, αν, θέλουμε να προβάλλουμε κάποια ένσταση, αυτό έχει τεθεί υπόψη μας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που θέτουν τα μέλη της Επιτροπής μας. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρώπη, τι προτίθεται να κάνει κάθε χώρα μέλος, τι υποδομές θα απαιτούνται, οι ε, κατασκευαστές έχουν έτοιμα τα μηχανήματα και ούτω καθεξής. Όλοι θέλουμε καλές οδικές συνθήκες κυκλοφορίας. Όλοι θέλουμε ταχεία ε, παροχή υπηρεσιών διάσωσης εφόσον απαιτείται και να διευκολύνονται αυτά εφόσον κάποιος υποστεί ένα τύχημα, αλλά κύριε Πρόεδρε δεν έχουμε ενημέρωση και είδα οι συνάδελφοί μου, κυρία Μάσιν και άλλοι, έθεσαν το θέμα. Πού κινούνται τα πράγματα αυτά. Άλλωστε το e-call δεν το έχουν δεχτεί όλες οι χώρες, όχι επειδή απαραίτητα δεν θέλουν να βελτιώσουν τις τροχές συνθήκες, αλλά ίσως θεωρούν ότι υπάρχουν θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Δεν γνωρίζουμε καν προς τα που κινείται όλο αυτό. Και μέχρι τις 21 θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα καταθέσουμε πρόταση ψηφίσματος. Αυτό μου φαίνεται απαράδεκτο. Προτείνω να έχουμε τη δυνατότητα να το ξανασυζητήσουμε, να το συζητήσουμε περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, και να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει. Η 21η είναι δική μας ημερομηνία, όχι της Κομισιόν, έτσι, 21η Δεκεμβρίου, για να παραμείνουμε εντός χρονοδιαγράμματος. Η Κομισιόν επιθυμεί να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως έχουμε όλοι ε, θα έχουν, μάλλον θα καθησυχαστούν τα μέλη όταν ακούσουν ότι θα έχουν το χρόνο να δουν την πρόταση. Δεν είναι μια εκτεταμένη πρόταση όπου έχουμε αλλάξει τις τεχνικές προδιαγραφές των όσων θα πρέπει να ενσωματωθούν στο οχήματα. Του τρόπο με του οποίου οι δημόσιε υπηρεσίε οργανώνονται στα κρατη για να χειρίζονται τα επίγοντα τηλεφωνήματα αφορά ένα σύνολο απλών προδιαγραφών για το τι είδο στοιχεία χρειάζεται το σημείο απάντησης δημόσιας ασφάλειας για να μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά και να δρομολογήσει και να διαδώσει ε, μηνύματα επίγουσας ανάγκης. Ε, για να σας το εξηγήσω πιο απλά. Δηλαδή, αναμένεται να εφαρμοστούν όλα αυτά όταν θα έχουμε προτείνει το σχέδιο νομοθεσίας και πάλι θα είναι ένα σχέδιο οδηγίας μάλλον που θα ε, προσπαθήσει να καθοδηγήσει τα κρατημέλη όσον αφορά τι είδη μέτρων θα πρέπει να λεφθούν ώστε να οργανωθούν εθνικά τα σημεία επίγουσας ανάγκης. Όπως είπα σε εθνικό επίπεδο και όλα αυτά με μεγάλη ευελιξία διότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι υπηρεσίες αυτές από το ένα κράτος στο άλλο ενδιαφέρει. Επαναλαμβάνω ότι εδώ εμείς ακολουθούμε αυστηρά την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκφράστηκε με πολλές λεπτομέρειες και σαφήνεια στην έκθεση που έχετε υιοθετήσει. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Είναι μια πρώτη, ένα πρώτο σημείο, ένα πρώτο κομμάτι από αυτά που χρειάζονται. Και βεβαίως μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε περαιτέρω. και σε διαμερθωρητική μορφή. Ακόμα και διμερώς, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε για να σας απαντήσουμε σε όλα τα τεχνικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω αυτά που είπα. Αν κάποιος η ομάδα ε, θέλει να καταθέσει πρόταση κατά της υιοθέτηση της πράξης, θα πρέπει να το κάνει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Αν ομάδα ή κάποιος θέλει να παρατείνει τους δύο μήνες, τους τέσσερις μήνες θα πρέπει να στραφεί στους συντονιστές ώστε οι συντονιστές να αποφασίσουν αν το δέχονται ή όχι. Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ για την προσφορά αυτή, ότι μπορούμε να συναντηθούμε και δημερώς και να συζητήσουμε διάφορα θέματα, αλλά πιστεύω πως θα ήταν ενδιαφέρον και για τους υπολείπους συναδέλφους να ακούσουν τα επιχειρήματα. Γι' αυτό δεν είμαι πολύ ευτυχής να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα εκτός της Επιτροπής, διότι υπάρχουν κάποιες απόψεις άλλων κρατών μελών, τις οποίες απλώς δεν γνωρίζω. Εγώ θα ήθελα, θα προτιμούσα να έχουμε αυτή τη συζήτηση για κάποιες παρατηρήσεις κρίσιμες στην Επιτροπή μας και όχι σε έξτρα συνεδριάσεις, γιατί εμένα με ενδιαφέρει και η Λιθιονία, με ενδιαφέρει και η Ιταλία και δεν με ενδιαφέρει μόνο η Αυστρία. Γι' αυτό είμαι κάπως αμήχανη ως προς αυτή την προσέγγιση. Σαιντ; Εγώ φυσικά δεν είμαι εδώ εξ Επιτροπής. Απλώς άκουσα από την Κομισιόν και νομίζω πως είναι σαφές και στο κείμενο πως πρόκειται για θέματα που δεν είναι επίμαχα Δηλαδή δεν είναι τα επίμαχα θέματα που εσείς αναφέρατε. Αυτά θα έρθουν αργότερα όταν θα έρθει και το σχέδιο πρότασης στον επόμενο χρόνο. Και φυσικά και θα συζητηθεί στην Επιτροπή το θέμα αυτό. Το θέμα που εμείς πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν είναι αν αυτό το καθαρά τεχνικό, τα τεχνικά ζητήματα, πώς θα πρέπει να τα εξετάσει η Επιτροπή μας, είμαστε κατά ή όχι και αν όχι αν έχουμε αρκετό χρόνο για να το εξετάσουμε στις επόμενες δύο εβδομάδες. Και η Κομισιόν είναι πρόθυμη να επανέλθει είτε σε διμερές επίπεδο είτε στους συντονιστές τους όπου θέλουμε. Εγώ προσωπικά ε, ε, θα κοιτάξω πιο προσεκτικά το κείμενο και εάν το θεωρήσω απαραίτητο να έχω περισσότερες πληροφορίες θα το ζητήσω να ε, Πανέλθουν ή να επανέλθουν στους συντονιστές. Αξίζει να διαβάσετε το κείμενο, ναι. Παρακαλώ, λοιπόν, διαβάστε το κείμενο. Είναι μόλις το 1 τρίτο του μεγαλύτερου φακέλου των εφιών συστημάτων μεταφορών. Πριν να βουτήξουμε λοιπόν και να πούμε δεν έχουμε χρόνο κτλ. Διαβάστε το το κείμενο και μετά φυσικά έχετε τα δικαιώματά σας όπως σας τα περιέγραψα για να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνουμε ως κοινοβούλιο. Το σημείο αυτό θα το βάλουμε στην ατζέντα, ώστε όλοι από τη Λιθουανία στην Ελλάδα να μπορούν να έρθουν και να ακούσουν τη συζήτηση. Το βάλαμε στην ατζέντα και εδώ είμαστε, ορίστε, τρεις και ο κούκος και ένα σωρό άδεια έδρανα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σα είπα ποια είναι η διαδικασία, τώρα εξαρτάται από εσά. Ευχαριστώ την Κομισιόν και τώρα αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών.